Sorry παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας. Μπορεί να είμαστε μόνο δύο μέλη παρόντα, αλλά ας ξεκινήσουμε. Ξεκινούμε με μια μικρή αλλαγή ε, από τη χθεσινή μερίσια διάταξη. Θα ξεκινήσουμε το σημείο 10, την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας σε μέσα πληρωμών πλήν των μετρητών. Θα μας κάνει την παρουσίαση η συγκέντρια κυρία Σιλβή Ιβόν Κάουφμαν. Θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής της. Λυπάμαι που χρειάστηκε να περιμένει τόση ώρα, Σιλβία. Έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλή σας μέρα. Σε όλους τους συναδελφούς και τις συναδελφούς. Ζούμε σε καιρούς με ραγδαίες αλλαγές κυρίως λόγω της ψηφιοποίησης και αυτό έχει επιπτώσεις και στον τρόπο με τον οποίο πληρώνουμε ε, με πιστωτικές κάρτες, ε, εμβάσματα διαδικτυακά, ακόμα και με εικονικά νομίσματα, πάντως χωρίς μετρητά. Όλα αυτά ε, αυξάνονται και αυτό ταυτόχρονα προσελκύει εγκληματίες. Έχουμε στοιχεία από το 2013 όπου η απάτη με πιστοτικές κάρτες στην Ευρώπη προκάλεσε ζημία τουλάχιστον ε, 1,44 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό μάλλον, από ό,τι φαίνεται, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πανευρωπαϊκές στατιστικές για απάτες γενικά με, μέσα πληρωμής διαφορετικά από τα μετρητά. Ε, το διαδίκτυο η απάτη έχει συχνά διασυνοριακή διάσταση. Οι δράστες και τα θύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται στην ίδια χώρα και αυτό προφανώς δυσκολεύει τις διοκτικές αρχές ε, στις έρευνες οι αξιόπινες πράξεις, ε, η διάρκεια ε, τέλους του εγκλήματος ε, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στόχος της οδηγίας είναι να έχουμε προδιαγραφές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάταξη να χαρακτηρίζεται κακούργημα το αδίκημα αυτό και πραγματικά αξίζει να υποστηριχθεί. Ήδη έχουμε ρύθμιση, μια απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου του έτους 2001, αλλά οι κανόνες της εποχής ε, προφανώ δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα, αρκεί μόνο να σκεφτεί κανείς ε, τις τεχνολογικές εξέλιξεις. Ε, στη μελέτη αντικτύπου και στην πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρκετά θετικά επιχειρήματα για αναθεώρηση των σημερινών διατάξεων. Προτείνει κάποιες αλλαγές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μεταξύ άλλων αφορούν διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των ε, συναλλαγών με εικονικά νομίσματα, ε, ε, εξίσωση των κακοργημάτων, ιδιαίτερα στην απάτη στο διαδίκτυο και κατώτατες ποινές και κύρωσης. Επίσης, γίνεται σαφής λόγος για τη δικαιοδοσία ε, γενικά ε, και για τα θύματα βέβαια κάποιες πρόνοιες είναι πολύ καλή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η βελτιωμένη διασυνοριακή συνεργασία των διοκτικών αρχών είναι στοιχειώδης για τη δίωξη κακουργημάτων και εγκλημάτων που δεν γνωρίζουν πια ε, σύνορα. Διευκολύνεται και η δήλωση και η καταγραφή τέτοιων απατών και βελτιώνονται οι στατιστικές. Επίσης, υποστηρίζω την ε, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταθέσει νέα νομοθετική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα στα πλαίσια ε, της εναρμόνισης με τη συνθήκη της Λισαβόνας και στο ποινικό δίκαιο που είναι συνομοθέτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παίζει σημαντικό ρόλο. Ως εισηγήτρια λοιπόν θα ήθελα να συμπληρώσω και να ενισχύσω περαιτέρω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξού και έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες. Να σας αναφέρω πέντε από αυτές. Πρώτον, ενισχυμένη υποστήριξη των θυμάτων. Γιατί όποιος έχει πληγεί από απάτη με πιστοτικές κάρτες, εφίσταται τις συνέπειες και στη συνέχεια. ο απατεώνας ε, χρησιμοποιεί την ταυτότητα του θύματος και αυτό μπορεί να πλήξει όχι μόνο τη φήμη του αλλά και την ε, πιστοληπτική του δυνατότητα και ικανότητα. Ε, αυτό μπορεί να καταπολεμηθεί και με πιο αξιόπιστα συστήματα δήλωσης διαδικτυακά της απάτης. Δεύτερον, η Eurojust και η Europol θα πρέπει όσο γίνεται να συμμετέχουν περισσότερα έτσι ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Στη συνέχεια, πρόληψη των αξιόπινων πράξεων αυτών είναι πάρα πολύ σημαντική. Ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες θα πρέπει ο καταναλωτής να έχει στα χέρια του σύμβουλες και χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορεί να θωρακιστεί ε, κατά της απάτης της διαδικτυακής. Επειδή υπάρχει επίσης εδώ πεδίο δράσης, που είναι αναγκαίο θα πρέπει να μειωθεί η προθεσμία που έχουν τα κράτη-μέλη για να μεταφέρουν στο εθνικό του δίκαιο την οδηγία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεωθεί μετά από μια τέτρα τετραετία να κάνει αξιολόγηση τη εφαρμογή τη οδηγία. Πρόεδρε, τελειώνοντα αν μου επιτρέπετε μια πολύ σημαντική παρατήρηση κατά τη γνώμη μου. Στο άρθρο 2 της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται κάποιοι ορισμοί και μάλιστα όλοι οι ορισμοί που έχουν σημασία για τη συγκεκριμένη οδηγία. Αλλά για να είμαστε συνεπείς ε, και με την υπόλοιπη νομοθεσία συνεννοηθήκαμε με την Επιτροπή που κανονικά ε, θα ήταν αρμόδια ε, επί της Συνεννοηθήκαμε λοιπόν να μην κάνουμε εμείς εδώ στη ΛΥΒΕ τροπολογίες για το άρθρο 2, να μην δεχτούμε τέτοιες τροπολογίες να πάρουμε τις, τους ορισμούς από την οδηγία ε, για την ομοποιήση εξόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δηλαδή στο άρθρο 2 να αντιγραφούν οι ορισμοί από την άλλη οδηγία όπως έχουν χωρίς καμία τροποποίηση. Για τις ε, προθεσμίες τώρα και το χρονοδιάγραμμα. Ε, προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών λίγη στις 11 Απριλίου, στις 5 ώρα το απόγευμα θα ψηφίσουμε, ε, μάλλον θα συζητήσουμε 25 και 26 Απριλίου εδώ στην Επιτροπή μας της τροπολογίας και αν όλα πάνε καλά προβλέπεται ψηφοφορία στις 25 Ιουνίου στην Επιτροπή μας. Αυτά Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. ευχαριστούμε Σίλβια Για το τελευταίο σχόλιο σου το διαδικαστικό να διευκρινίσω ότι το άρθρο 2 της, ε, της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εμπίπτει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό των διαφόρων μέσων πληρωμής, ας μην ξεχνούμε ότι οι τροπολογίες για το άρθρο 2 δεν θα ψηφιστούν στην δική μα Επιτροπή, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, γιατί παραλαμβάνουν θέματα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Και μα είπε και για τι προθεσμίε. Υπάρχουν σχόλια από του και ο κύριος Μέλο. Ευχαριστώ. Ε, επιγραμματικά. Συμφωνούμε με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την κρίνουμε πολύ σημαντική για το διευρυμένο πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας. Επίσης, συγχαίρουμε την εισηγήτρια για την πρότασή της ε, ασθενιζόμαστε τις απόψεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πράσπιση των μηχανισμών που διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για ε, εγκλήματα που έχουν τελεστεί μεταξύ των αρμόδιων αρχών και προσδιορίζει τι αρμοδιότητες της Eurojust και της Ευρωπόλ σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και επίσης προτείνει συντομότερε προθεσμίες για την μεταγραφή της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Ε, μπράβο σας. Ε, θα σας στηρίξουμε στην προσπάθειά σας και επίσης θα καταθέσουμε τροπολογίες που ελπίζουμε να κριθούν ε, εύστοχες και δόκιμες από την εισηγήτρια και να συμπεριληφθούν στο κείμενό της. Ευχαριστώ κύριε Ζολή. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την ε, Σιλβί Καφμάν για την έκθεση της. Πολύ καλή εξαιρετική θα έλεγα βάση για τις περαιτέρω εργασίες και η οδηγία είναι πολύ σημαντική για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τις απάτες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η προηγούμενη απόφαση πλαίσιο δεν αυθυγραμμιζόταν ε, με τις πολύ ε, ραγδαίες εξέλιξεις στα μέσα, εικονικά κυρίως ψηφιακά μέσα πληρωμών. Οπότε ήταν ώρα για αναθεώρηση της προηγούμενης θέσης και είμαι υπέρ μιας ε, ε, πιο μεγάλης εμπλοκής της ε, Ευρωπόλ και της Eurojust και μεγαλύτερη προστασία των θυμάτων. Και πολύ εύστοχα επισημαίνεται ότι είναι πολύ ενοχλητική αυτή η κατάσταση και ταλανίζει το θύμα που είναι θύμα συμφεταρισμού ταυτότητας για πάρα πολλά χρόνια μετά την διάπραξη του εγκλήματο. Επίση η ιδέα τη απλούστευση των συστημάτων προσφυγής και τη θέσπιση ενός ε, διαδικτυακού συστήματος επιγραμμικού για τις, κοιν... τις, ε, τις κοινοποίησεις ε, των εγκλημάτων, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά κάποια σημεία χρήζουν περαιτέρω διευκρίνησης. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να προτείνουμε την σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Τμήματος πληροφορι... οικονομικών πληροφοριών. Θα ήταν πολύ ε, δόκιμο να γίνει ένα τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τι υποθεσμίε για την ε, επισήμαση ε, ή την, το, το συναγερμό, πολύ σωστά να συντομεύσουν και θα καταθέσουμε και εμεί τροπολογίε στο σχέδιο έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κοράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, δουλειά της, αλλά και την Επιτροπή για την πρόταση. Τι συμμεριζόμαστε. Όπως άλλωστε συμμεριζόμαστε και τις παρατηρήσεις της κυρίας Κάουφμαν. Ξέρουμε πόσο σημαντικό μέρος εσόδων για τις ε, κλιματικές οργανώσεις ε, αντιστοιχεί σε αυτές τις απάτες και γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ε, πρόκειται σε τελευταία ανάλυση για αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και πρέπει να το πλήξουμε το οργανωμένο έγκλημα εκεί ακριβώς όπου πουνάει δηλαδή στα έσοδα στο οικονομικό σκέλος και νομίζω ότι αυτό είναι και το κύριο κομμάτι της δουλειάς που έχω κάνει και εγώ στην οδηγία κατά της ε, ανακύκλωσης παρανομών εσόδων. Για το σχέδιο εκθέσης, όπως είπα, σύμφωνα με πολλά σημεία της και κυρίως δύο κομμάτια που και εγώ θεωρώ πολύ σημαντικά. Την έμφαση που δίνεται στο θύμα, στα θύματα και την ε, προσπάθεια για περισσότερη φροντίδα και προστασία για αυτά, αλλά ταυτόχρονα και στο σκέλος που έχει να κάνει με τη διευκόλυνση των καταγγελιών, συστήματα online επί παραδείγματι που αναφέρονται για την καταγγελία των απατών. Η περίοδος μεταφοράς ε, στο εθνικό δίκαιο μειώνεται από τους 24 στους 12 μήνες και σε αυτό συμφωνώ επίσης. Μια σειρά θεμάτων ε, από την πρόταση της Επιτροπής με ενδιαφέρουν και πρόκειται να καταθέσω σχετικές τροπολογίες. Ε, στα θέματα της απομίμησης ε, πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί, πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση των μέτρων. Τα μέτρα, παραδείγματι, για την επίλυση των αρνητικών συγκρούσεων δικαιοδοσίας, όταν δηλαδή καμία αρχή δεν θεωρεί ε, αυτήν αρμόδια και άρα δεν γίνεται δίωξη του εγκλήματος. Θα ήταν καλό να υπάρχει μια λύση μέσω της Eurotest ενδεχομένω και με την ε, επιβολή ιεραρχικά μιας ε, λύσης, δηλαδή ορισμό άνωθεν του ποια θα είναι η αρχή, η δικαιοδοτική που θα πρέπει να ασχοληθεί με την υπόθεση για να αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις αρνητικής δοσηδικίας. Αυτά και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που να μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ τους Κιώδης. Ο κύριο Τσικόφσκι έχει πει στο λόγο. Ευχαριστώ Κλοντ και ευχαριστώ Σίλβια για την παρουσίαση και την εξαιρετική δουλειά. Θα πρότεινα να κάνω και έχω κάποιες ε, τροπολογίες συγκεκριμένες για συγκεκριμένα θέματα. Ε, ουσιαστικά για να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα ώστε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι Συμφωνώ πάντως με το κείμενό σου απολύτως και χαίρομαι που ορίζεις και την ευθύνη που ε, ε, υπάρχουν τα κράτη στο να προσφέρουν ε, υποστήριξη στα θύματα. Και ιδιαίτερα βέβαια μας ενδιαφέρει η προστασία των εγκλημάτων αυτών των οργανωμένων μορφών εγκλήματος. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την έκθεση και ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σίλβη. όπως βλέπεις ε, πολύ θετική ανταπόκριση των συναδέλφων. Θέλεις κάποια τελικά σχόλια? Ναι, πολύ σύντομα Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ τους συναδέλφους. Χαίρομαι ιδιαίτερω ε, για την αναφορά στο ζήτημα της προστασίας των θυμάτων που αναφέρατε και εσείς, γιατί για το Κοινοβούλιο πρόκειται για ένα κεντρική σημασία ζήτημα όπως και το ζήτημα της ε, ιεράρχησης των αρμοδιοτήτων, του να είναι σαφές ε, ποιος είναι αρμόδιος στο θέμα της δικαιοδοσίας και η παραπομπή η συμμετοχή στη διαδικασία της Eurojust ώστε να υπάρχουν σαφείς δυνατότητες για τη λήψη των αποφάσεων, να μην έχουμε ούτε ε, θετική ούτε αρνητική σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών και των αρχών τους. Χαίρομαι ιδιαίτερως, περιμένω τις ε, τροπολογίες με χαρά και είμαι βεβαία ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία που θα οδηγήσει σε ένα καλό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Επομένω Ιβόν, ε, και μια και θέλει και η Επιτροπή το λόγο, αν δεν έχει αντίρρηση, παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ. Όντως, πολύ λακωνικά χαιρετίζουμε την, το σχέδιο έκθεσης και ιδιαίτερα τις τροπολογίες που ενισχύουν την αρρωγή προς τα θύματα. Πολύ αξιόλογες προτάσεις μας. Προβληματίζουν κάπως οι τροπολογίες που προβλέπουν υποχρεωτική ενημέρωση για τα φαινόμενα απάτης. Στη μελέτη επιπτώσεων το εξετάσαμε και οι ενδιαφερόμενοι και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα θεωρούν ότι ε, είναι υπερβολική επιβάρυνση και των δικαστικών αρχών και του κλάδου και ε, το πλεονέκτημα δεν είναι ιδιαίτερο από μια τέτοια υποχρεωτική υποβολή αναφοράς. Προτιμούμε μια ε, τεχνολογικά ουδέτερη οδηγία που ε, εξασφαλίσει το απαραίτητο πλαίσιο στις ε, δικαστικές και αρχές επιβολής του νόμου για να μπορούν να εφαρμόσουν την οδηγία προσαρμοσμένη και στις νέες τεχνολογικές εξέλιξεις. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε την εισηγήτρια για το έργο της. Η προθεσμία, όπως είπε και η συγγετρία για τις τροπολογίες, λήγει στις 11 Απριλίου στις 5 το απόγευμα. Κανονικά τώρα πρέπει να περάσουμε στο σημείο 11, αλλά περιμένουμε ακόμη το διευθυντή της Frontex, τον κύριο Λετζέρη, που κανονικά αναμένεται για τις 10 ε, δεν έχει έρθει ακόμη. Colleagues, if you don't mind, if we could um, have a short pause until 9.40. Οπότε θα κάνουμε μια μικρή διακοπή μέχρι τις 10 παρατέταρτο και θα περάσουμε τότε στο σημείο 11 για τη Frontex. Παρακαλώ επιστρέψτε 10 παρατέταρτο.

Δεν προσθέτουμε μουσική υπόκριση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών μονίμως, αλλά επί δυστυχώς δεν ακούγεται το μικρόφωνο του. Α, εντάξει. Και όμως ήταν πολύ καταπρέντικη η μουσική αυτή η υπόκρουση. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για την, την υπομονή που δείξετε. Ο κύριος Λεζερή έχει ήδη ε, έρθει και η κυρία Φερνάντες, η υπεύθυνη θεμελιωδών δικαιωμάτων του Frontex, ε, επίσης είναι εδώ και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα θα γίνει μια παρουσίαση ε, βίντεο, εξού και η μουσική που ακούσατε πριν από λίγο, μια σύντομη παρουσίαση από βίντεο. Μετά θα ακούσουμε τον κύριο Λεζερή που θα μας παρουσιάσει την επιχείρηση Θέμης θα μας ενημερώσει για την επιχείρηση αυτή. Αλλά φυσικά στη συνέχεια μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για το Frontex και για, την, ε, ε, ε τον Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Επίσης, συντονιστέ συντονιστές να καλέσουμε και την υπεύθυνη θεμελιωδών δικαιωμάτων του Frontex, του οργανισμού Frontex, την κυρία Φερνάντες, για να μας ενημερώσει Οπότε μετά τον κύριο Λεζερή θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση και η κυρία Φερνάντες και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Είναι μια προσθήκη στην τακτική ενημέρωση που μας κάνει κανονικά ο κύριος Λεζερή. Μια σύντομη εισαγωγή και μετά θα περάσουμε στα θέματα ουσίας. Κύριε Λαζαρή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σας αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Παρακολουθήσατε το βιντεάκι που συνοψίζει ουσιαστικά τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης Θέμης. Καταρχήν να δούμε τις επαρχές αυτής της επιχείρησης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι συνεργαστήκαμε με τα κράτη-μέλη και κυρίως με τις Ιταλικές αρχές. Ε, ξεκινήσαμε το καλοκαίρι του 2017 την επιχείρηση αυτή μετά από αίτημα της Ιταλίας αλλά και τα δικά μας πορίσματα έδειξαν ότι κάποιες μορφές συμπεριφοράς ε, της μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος άλλαζαν στη Μεσόγειο. Είχαμε περισσότερες ροέ από την Τινησία Αλγερία, άμεσε ε, ροέ από την Τουρκία στην Ιταλία και από την Ελλάδα προ την Ιταλία. Περισσότερες απειλέ ε, ασφάλειας, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, καθώς και δυνητικές τρομοκρατικές απειλέ λόγω ε, αφήξεων που πέρασαν απαρατήρητες και γνωρίζετε και για την κατάσταση του ΝΤΕΣ, του Ισλαμικού κράτους στη Συρία και το Ιράκ. Την 1η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους η επιχείρηση Θέμης εγγενιάστηκε και επίσημα και υπάρχει εδώ ένα μείγμα συνέχισης και επιβολής ε, νέων ε, ε, ιδεών. Καταρχήν, ως προς τη συνέχεια με την προηγούμενη επιχείρηση, τον Τρίτονα. Καταρχήν, ε, έρευνες και διάσωση στη θάλασσα είναι και αυτό το και των στόχων της νέας επιχείρησης της Θέμης. Ε, μάλιστα, οι προσπάθειές μας στηρίζουν το, συστημ το κέντρο θαλάσσιας διάσωσης και χωρίς περιορισμό μάλλον. Δηλαδή, η εμβέλειά μας η επιχειρησιακή δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην έρευνα και διάσωση. Επίσης, ε, αναπτυσσόμαστε και στα κέντρα καταγραφής ε, στην Ιταλία, δηλαδή στα χερσαία κέντρα καταγραφής, ε, προκειμένου να βοηθήσουμε την Ιταλία να ενημερώσει τους μετανάστες, να συγκεντρώσει τα κτηλικά αποτυπώματα και τα πιο ευάλωτα άτομα να τα παραπέμψει προς το Γραφείο για τη Μετανάστευση και τις αρμόδιες αρχές ασύλου. σε, σε ε, ε, ελέγχους ασφάλειας της δεύτερης γραμμής που γίνονται από, την, από τις τελικές αρχές σε περίπτωση, και την Γεροπόλη σε περίπτωση που έχουμε κάποιες ε, υπόνοιες ε, ή αμφιβολίες για τα θέματα ασφάλειας. Επίσης έχουμε ε, στενή συνεργασία με τη UNAFORMED, την επιχείρηση Σοφία της UNAFORMED από τις αρχές του 2015 που ισχύει. Αυτά είναι τα στοιχεία της συνέχειας σε σχέση με προηγούμενες επιχειρήσεις. Τώρα, οι νέες πτυχές ε, της επιχείρησης ε, Θέμης. Ποιες είναι. Καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι ε, έχουμε κάποιες λειτουργίες και άκτο φυλακής με βάση τη νέα μας εντολή και χρησιμοποιούμε τα διδάγματα από το πιλωτικό πρόγραμμα των επιχειρήσεων ακτοφυλακής του 2017 και έτσι αναπτύξαμε ένα πιο, μια πιο στιβαρή προσέγγιση για τις της ακτοφυλακής με προσανατολισμό σε θέματα επιβολής νόμου παράλληλα με τα, τα καθήκοντά μας για έρευνα και διάσωση. Να σας υπενθυμίσω ότι πέρυσι περίπου 800 ανταλλαγές είχαμε με την ΕΦΚΑ σε ό,τι αφορά ύποπτα σκάφη και έπτα περιπτώσεις ε, ρήπασης που διερευνήσαμε με την ΕΜΣΑ πέρυσι, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Και αντλήσαμε κάποια διδάγματα σε σχέση με το πιλωτικό πρόγραμμα και τη δημιουργία ικανοτήτων των λειτουργιών ακτοφυλακής. Επίσης, ε, αξιοποιήσαμε την εμπειρία μας ε, σε ό,τι αφορά την επιβολή του νόμου σε θέματα καταπολέμησης λαθρεμπορή ναρκωτικών στην, στην επικράτη Ιταλίας, Αλβανίας και Ελλάδας. Και επικεντρώσαμε τις δραστηριότητες επιβολής του νόμου και ασφάλεια αυτή την ευρύτερη περιοχή. Η επιχείρηση Θέμης ε, ε, χρησιμοποίησε κάποια διδάγματα του, του νέου επίπεδου χώρου επιτήρησης ε, που αυτόνομα πια εξασφαλίζουμε με τα δικά μας αεροσκάφη και καταφέραμε να εντοπίσουμε ε, αυτόν τον αέριο χώρο, ε, στον αέριο αυτό χώρο κάποιες αδυναμίες, κάποια κενά που μέχρι στιγμής είχαν περάσει απαρατήρητα. Ε, για παράδειγμα, κάποιες ε, ε, ροές μετανάστευσης που δεν είχαν εντοπιστεί κυρίως από Αλγερία και την Ισία, κάποια προβλήματα προς την ασφάλεια λόγω αυτών των ε, παράνομων και ασυνήθιστων ροών που πέρασαν παρατήρητες ε, εισήλθαν από την Αλγερία και την Τινησία προς την Ευρώπη και επίσης κάποιες άλλες δραστηριότητες όπως παράνομη αλία ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Επίσης αναπτύξαμε ε, στα πλαίσια της επιχείρησης θέμης κάποιες εσωτερικές μορφές ε, επιτήρησης, κάποια φορτηγά θερμο, ε, θερμοπτικής ε, τεχνολογίας και έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιους μετανάστες που φτάνουν στο, στην Ιταλική επικράτεια και προηγουμένως δεν είχαν εντοπιστεί. Επίσης τροποποίησαμε την επιχειρησιακή μας εμβέλεια το επιχειρησιακό πεδίο εφαρμογή μας ε, σε συνδυασμό συνεργασία με τι τελικέ αρχέ. Με βάση τον κανονισμό, ο εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού υπογράφει το επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά θα πρέπει να φροντίζει ότι το, η, τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών τη χώρα υποδοχή, δηλαδή τη Ιταλία προκειμένου. Οπότε επεκτείναμε τον επιχειρησιακό μα χώρο από τα δυτικά τη Αρδινία μέχρι την Αδριατική μπροστά δηλαδή στα Δυτικά Βαλκάνια και με αίτημα των Ιταλικών αρχών ο επιχειρησιακός μας χώρος δεν επικαλύπτει ή δεν συμπίπτει με τη δηλωμένη μαλτέζικη ζώνη έρευνας και διάσωσης και μετά από αίτημα της Ιταλίας δεν συμπίπτει ούτε με τη δεδηλωμένη ε, λιβική ζώνη έρευνας και διάσωσης γιατί πέρυσι το καλοκαίρι θυμάστε ε, δηλώθηκε ε, μια λιβική τέτοια ζώνη έρευνα και διάσωση. Εμείς αποφεύγουμε τις επικαλύψεις με αυτές τις περιοχές. Η επιχείρηση Θέμη αξιοποίησε και τα διδάγματα που αντλήσαμε κατά την εφαρμογή της συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων. Θα θυμάστε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο Frontex, μπορεί πλέον να συγκεντρώνει και προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια κάποιων ε, δραστηριοτήτων debriefing στα εξωτερικά σύνορα. Οπότε συγκεντρώνουμε, επεξεργαζόμαστε και ε, ανταλλάσσουμε προσωπικά δεδομένα για ε, διερευνήσεις ποινικών αδικημάτων και με τα κρατημέλη και με την Ευρωπόλ που είναι ο κύριος εταίρος μας σε θέματα τέτοια. Έτσι σταδιακά φτάσαμε στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο, στη νέα επιχείρηση, την επιχείρηση Θέμης και αλλάξαμε και το όνομα. Το όνομα Θέμης ε, αντικατοπτρίζει καλύτερα την αισθήση της ε, επιχείρησης αυτής σε επιβολή του νόμου, γιατί η Θέμης είναι η θέα της δικαιοσύνης, θεότητα της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου. Και μάλιστα ταυτόχρονα αναπτύξαμε και τις λειτουργίες μας σε θέματα ακτοφυλακής και ε, συμμετέχουμε ενεργά και αποτελεσματικά στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Τώρα κάποια συμπεράσματα και ποια είναι η κατάσταση φέτος. Καταρχήν θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είναι σαφές ότι το επιχειρησιακό σχέδιο το διευκρινίζει ότι μετά από τρίμηνη εφαρμογή της επιχείρησης θέμης θα γίνει μια αξιολόγηση. Οι Ιταλικές Αρχές και ο Frontex συμφώνησαν στην ανάγκη να μην περιμένουμε έναν χρόνο ολόκληρο, αλλά να γίνει πρώτη αξιολόγηση μετά από το πρώτο τρίμηνο. Δηλαδή αρχές ε, ε Μαΐου, τέλη Απριλίου θα ε, διενεργήσουμε αξιολόγηση από με τις Ιταλικές Αρχές. Φέτος από την 1η Ιανουαρίου είχαμε περίπου 6.000 ε, παράτυπους μετανάστες που εντοπίσαμε στην Κεντρική Μεσόγειο, δηλαδή μίαν, κατά 62% λιγότερο σε σχέση από πέρυσι. Η Λιβύη, και αυτό είναι ενδιαφέρουσα εξέλιξη, η Λιβύη είναι η χώρα αναχώρησης μόνο στο 71% των περιπτώσεων. Πέρυσι ήταν πάνω από το 95% των περιπτώσεων οι, η από τη Λιβύη. Πού έγινε η διαφορά τώρα. Το 20% των αναχωρήσεων ε, ε, προέρχονται από την Τινησία και η Τουρκία ή μάλλον οι άμεσε ε, ε, από την Τουρκία ήταν 5%, από την Αλγερία 2% και θαλάσσια από την Ελλάδα προς την Ιταλία 2% των αναχωρήσεων. Και μάλιστα σε μία περίπτωση ε, είχαμε προέλευση το Μαυροβούνιο και είναι πολύ νωρίς να, διαπιστώσουμε αν είναι μια προσπάθεια διάνοιξης νέου διαδρόμου ήταν τυχαίο και έκτατο αυτό. Yeah, δεν ξέρουμε αν δημιουργείται νέα, νέα διαδρομή από τα Δυτικά Βαλκάνια προς την εδοχώρα της ε, ή προς την υπηρετική μάλλον Ιταλία. Τώρα προς τις εθνικότητες των μεταναστών, η πρώτη εθνικότητα φυσικά είναι η Ερυθρέα, Κάτοικη της Ερυθρέας, πάνω από 1500 φέτος. Και η δεύτερη εθνικότητα που φτάνει στην Ιταλία στα πλαίσια της επιχείρησης Θέμης είναι την ίση. Περίπου 1.200 την ίση κατέφτασε στην Ιταλία. Μετά η Νιγηρία, Πακιστάν, Λιβύη. Και αυτό είναι καινούριο. Έχουμε και από τη Λιβύη μετανάστες. Αυτή είναι μια νέα τάση. Και από την ακτή του Ελεφαντοστού. Τώρα, ως προς τα στοιχεία για την έρευνα και διάσωση από τις αρχές του 2018 ο Frontex συμμετείχε σε 23% των επιχειρήσεων ε, έρευνας και διάσωσης, δηλαδή ο αριθμός των περιπτώσεων ή των ε, διασωθέντων είναι το 23% της, συμμετοχή, της συμμετοχής μας και το ίδιο ακριβώς ποσοστό είχαμε και το 2017 και το 2017 η Frontex ε, διενήργησε το 23% των επιχειρήσεων, έρευνα και διάσωση. Δεν είναι αυτή η τελική αξιολόγηση και όπω σα είπα τέλη Απριλίου θα γίνει η κοινή αξιολόγηση με τι ιταλικέ αρχέ για την επιχείρησή μα. Καταρχήν ό,τι αφορά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, εκεί είχαμε μια πολύ, ε, ένα πολύ επιτυχή εντοπισμό πριν από τρει μέρε, 550 κιλά ναρκωτικών, μαριχουάνας κυρίως, εντοπίστηκαν από ένα αεροσκάφος που αναπτύξαμε στα πλαίσια του, ε, του Θέμης, της επιχείρησης Θέμης και έκανε περιπολία το αεροσκάφος κοντά στην Απουλία, δηλαδή νότιο-ανατολικά της Ιταλίας απέναντι στην Αλβανία και το αεροσκάφος αυτό εντόπισε ύποπτη συμπεριφορά και μετά από συντονισμό με τις Ιταλικές αρχές εντοπίστηκε αυτό το φορτίο, αυτή η παρτίδα και συνελήφθησαν μάλιστα και λαθρέμποροι ναρκωτικών. Εν κατακλείδη θα ήθελα να τονίσω ότι παρακολουθούμε εκ του και στην, τον αντίκτυπο της επιχείρησης θέμης σε θέματα έρευνας και διάσωσης και διαπιστώνουμε ότι η επιχείρηση αυτή, η ιδέα της επιχείρησης αυτής ε, εμπίπτει σε μια, στο περίπλοκο και είναι κατάλληλη για το περίπλοκο αυτό μεσογειακό περιβάλλον γιατί έχουμε νέες ε, διόδους από νέες χώρες αναχώρησης, ε, προέλευσης, την Ισία για παράδειγμα, αλλά δεν είναι η μόνη. Επίσης, είναι πολύ πιο ευέλικτες οργανωμένα, τα οργανωμένα κυκλώματα εγκλήματος και έχουμε διάφορους εγκληματικούς συνασπισμούς και συμμαχίες ε, που αφορούν και εμπορία ανθρώπων και λαθρεμπόριο ναρκωτικών και μερικές φορές εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες αυτά τα οργανωμένα κυκλώματα. Ακόμη και σε λαθρεμπόριο όπλων έχουν επεκταθεί. Οπότε είναι πολύ πιο ευέλικτα αυτά τα κυκλώματα και έχουμε λιγότερες ε, επιχειρήσει ε, ε, δράσεις, δραστηριότητες ελευθερεμπορίας που αφορούν ε, τις τελωνιακέ αρχές. Αυτό, το ελευθερεμπόριο αφορά περισσότερο ε, τα, τις δικές μας αρμοδιότητες, συνόρια φυλακής και ακτοφυλακής. Πάντως, όλοι έχουμε επίγνωση ότι και οι τρομοκρατικές απειλές και οι απειλές στην ασφάλεια δεν έχουν υποχωρήσει σε σχέση με πριν από μια διετία. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε οι παράνομες διελεύσεις να μην σχετίζονται με προβλήματα ή απειλές της ασφάλειας. Αυτά σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για τη συζήτηση, αλλά πρώτα να ακούσουμε την υπεύθυνη θεμελιωδών δικαιωμάτων και να μας παρουσιάσει τη δική της σκοπιά του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Yes, and just to explain to... Ναι, θα ήθελα να εξηγήσω στους συναδέλφους. Ζήτησαν οι συντονιστές να ακούσουμε και την κυρία Φερνάνδης να έρθει εδώ στη συνεδρίασή μας. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσετε στην Επιτροπή. Όχι, δεν είναι. Έχω ξανάρθει αλλά παλιά. Ναι, ναι, έχει πέρασει αρκετό χρόνο. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο και μετά θα γίνει συζήτηση. Thank you, Mr. Thanks a lot. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, αλλά και για την πρόσκληση που μου απευθύνετε να μιλήσω στα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθερίων και στο Κοινοβούλιο. Είναι πραγματικά τιμή για μένα να βρίσκομαι ενώπιό σας ως ε, σύμβουλος και ε, ανεξάρτητη ε, ε, στη Frontex. Μου ζήτησα να μιλήσω για τρία πράγματα. Πρώτον, ο μηχανισμός καταγγελιών και παραπώνων και πώς λειτουργεί. Ε, αυτό έχει γεννήσει μεγάλο ενδιαφέρον και στο Κοινοβούλιο εν ώψη του νέου κανονισμού ε, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Επίσης μου ζητήθηκε να μιλήσω για τα θεμελιώδη δικαιώματα τη επιχειρήσεις και για το, την επιχείρηση Θέμης. Αν μου επιτρέψετε με αυτή τη σειρά θα αναφερθώ στα θέματα. Ε, πρώτον, σε ό,τι αφορά το μηχανισμό καταγγελιών και παραγόντων, όπως είπα, τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2016 στο Frontex και έχει σχεδιαστεί ως μηχανισμός ελέγχου και παρακολούθησης για τα κατά πόσο συμμορφούνται προς ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οπότε πρόσωπα, ε, φυσικά πρόσωπα μπορούν να διαμαρτυρηθούν στον αρμόδιο ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις δραστηριότητε αυτές. Τι κάνουμε ελέγχουμε πρώτα το παραδεκτό ε, της καταγγελίας. Δεν ε, αφισβητούμε τα στοιχεία. Ε, βεβαίως είναι τυπική αυτή η διαδικασία για το κατά πόσο είναι παραδεκτή αυτή η καταγγελία. Όχι αν έγινε αυτή η δραστηριότητα στα πλαίσια των επιχειρήσεων του Frontex ή από τον ίδιο τον Frontex. και εξαρτάται ποιο είναι ο πάντα ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στην ε, αλληλογραφία, στην ανταλλαγή ε, των πληροφοριών και ο αρμόδιος για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο ίδιος εκτελεστικό διευθυντής ε, ελέγχει αυτές τις αναφορές, τις καταγγελίες και τις παραπέμπει σε εμάς για να δούμε αν θα δώσουμε συνέχεια ή αν θα κλείσουμε το θέμα. Υπήρξαν διάφορα ζητήματα ε, στην αρχή, ε, το πρώτο 18 μήνο. Ε, και έκτοτε έχουμε ένα αυτόματο σύστημα, μια, ένα έντυπο για τις καταγγελίες στην ιστοσελίδα μας που έχουμε συμφωνήσει με το Συμβουλευτικό Φόρουμ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Έχουμε και κανόνες που εγκρίθηκαν στη συνέχεια από τον εκτελεστικό διευθυντή και έχουμε αρχίσει και μια ε, καταγραφή, μια χαρτογράφηση ε, στις αρχές ε, των κρατών μελών που κατατίθεται αυτές οι αναφορές οι παραπέμπονται στα κράτη-μέλη, οργανισμούς θεμελιωδών δικαιωμάτων κλπ. Επίσης έχουμε διανύμει έντυπα και υλικό συνειδητοποίησης σε δέκα διαφορετικές γλώσσες. για να είναι πιο προσβάσιμος ο μηχανισμός. Όλα αυτά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Frontex. Επίσης, στην νέα ιστοσελίδα που θα ανανεωθεί προσεχώς θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγγελίας. Δεν χρειάζεται κάποιος να υπογράψει και να στείλει έντυπο, μπορεί να το κάνει και ηλεκτρονικά. Μέχρι τώρα Έχουμε 19 καταγγελίες ε, λάβει, 5 θεωρήθηκαν παραδεκτές και αφορούν ισχυρισμούς ε, παραβίασης του δικαιώματος στο άσυλο και της προστασίας ε, σε περίπτωση επιστροφής, απομάκρυνσης ή έκδοσης. Υπάρχουν και θέματα με ανηλίκους και έχουμε συμπεριλάβει και τα δικαιώματα των ανηλίκων. Τρεις από τις πέντε αυτές υποθέσεις καταγγελίες παραμένουν ανοιχτές και περιμένουμε να γνωμοδοτήσει ο αρμόδιος ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι αρχές των κρατών μελών. Και σε μία περίπτωση αποφασίστηκε να δοθεί συνέχεια ε, γραπτό σε συνεννόηση με τον εκτελεστικό διευθυντή. Ε, οι μη παραδεκτές καταγγελίες είχαν όλες να κάνουν με δραστηριότητες που δεν ήταν αυτές, αυτές εντός της εντολής του οργανισμού Frontex ή εντός του πεδίου δράσης. Αφορούσαν συνθήκες κράτησης, ε, ζητήματα ε, μέσων ενημέρωσης, εκκρεμούσες αποφάσεις για το άσυλο. Ο κόσμος έχει αγωνίες προφανώς και θεμητέ, και ρωτούσαν γιατί δεν έχει ληφθεί η απόφαση ή για τις τελικές αποφάσεις, για τις επιστροφές και προσφύγες, αλλά αυτά δεν είναι αρμοδιότητες ούτε του Frontex ούτε του ε, αρμοδίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση όλες οι καταγγελίες αυτές, οι παραδεκτές και μη ε, διαβιβάζονται στις αρμόδιες ε, κρατικές αρχές και στους διάφορους διαμεσολαβητές συνηγόρους του πολίτη, στα κράτη-μέλη, στους οργανισμούς που είναι γνωστό ότι έχουν τέτοιες δομές και ε, υποστηρίζουν τέτοιες ε, δράσεις. Εξορισμού εμείς ε, ελέγχουμε κατά, πόσο αυτές οι καταγγελίες έχουν σχέση με τη θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μεσολαβεί δικηγόρος. Μπορεί ο ίδιος ο διαμαρτυρός καταγγέλων να απευθύνεται σε εμά και εμείς τα ελέγχουμε. Και χαίρομαι για την υποστήριξη του Συμβουλευτικού Φόρουμ αναθεωρούνται τώρα οι κανόνες και σίγουρα στο μέλλον θα είναι σημαντική η συμμετοχή τους για τη διάδοση και προβολή του μηχανισμού. Πάρα πολύ κρίσιμο αυτό και πάρα πολύ χρήσιμο να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και που το έχουν ανάγκη πώς μπορούν να κάνουν καταγγελίες και τα παραπονά τους. Ε, για τη δεύτερη ερώτηση, το δεύτερο θέμα έρχομαι. Τι γίνεται με τα επιχειρησιακά ζητήματα. παρόλο που ήταν πολύ μικρή η προθεσμία, λάβαμε πολύ έγκαιρα τις εσωτερικές διαβουλεύσεις για όλες τις εκθέσεις. Ώρα που είμαστε μικρή ομάδα, λιγάριθμοι, εντός των χρονικών πλαισίων που έχουν συμφωνηθεί. Είναι πολύ σφιχτές οι προθεσμίες, αλλά προσπαθούμε να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα. Είναι πολύ χρονοβόρα αυτή η διαδικασία, αλλά σημαντική, γιατί προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ασφαλιστικές δικλείδες για να προστατεύουμε από παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης, μας έχει ζητηθεί να ε, ορίσουμε και στόχους για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων Και τώρα σε τεχνικό υπηρεσιακό επίπεδο προσπαθούμε να επεξεργαστούμε κάποιους δείκτες για να ε, μετρούν ε, τους στόχους και την, εγγύηση αμελιωδών δικαιωμάτων ε, στους τομείς όπου επιχείρει ο Frontex. Όπως είπε και ο εκτελεστικός διευθυντής για τα επιχειρησιακά σχέδια, προβλέπεται στον κανονισμό ο μηχανισμός παραπομπής Ε, σε περίπτωση που έχουμε θύματα δουλεμπορίου, τράφικ, ασυνόδευτους ανηλίκους, ε, ευάλωτες ομάδες ε, και άτομα που δικαιούνται διεθνούς προστασίας, πώς όλα αυτά να παραπέμπονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Έχει γίνει αυτό ήδη δύο φορές, πέρυσι μια φορά και μια φορά φέτος και είμαστε τώρα στο στάδιο της αξιολόγησης αν χρειάζεται διευκρίνηση, κάποια διαδικασία ή περαιτέρω ενημέρωση με συγκεκριμένα παραδείγματα. Επίσης, στα επιχειρησιακά σχέδια έχουμε και οδηγίες και εντολές και πληροφορίες σχετικά με το μηχανισμό κατακελιών για τον αρμοδίων, των αρμοδίων υπαλλήλων που πρέπει να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός. Ποια είναι τα προβλήματα. Καμιά φορά είναι η ίδια η διεθνής προστασία και πρόσβαση ερώτησης αυτή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους απάτριδες. Γι' αυτό έχουμε εκπονήσει ένα μέσο μαζί με την ΕΑΣΟ και ε, σε όλες τις ενημερώσεις ε, το αναφέρουμε αυτό. Ε, πιο πρόσφατα τώρα έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο να δίνουμε οδηγίες και κατευθύνσεις στα δικαιώματα των παιδιών, των ελικων σε θέματα φύλου ε, σε ειδικέ περιπτώσεις και ε, οδηγίες ε, στις ομάδες που επιχειρούν. Για τους ανηλίκους, πριν από αρκετό καιρό έχουμε έχουμε εντοπίσει στα αεροδρόμια τους ανηλίκους που χρειάζονται ειδική προστασία ε, στα κράτη-μέλη που βρίσκονται σε επικίνδυνες διαδρομές πάντα προς όφελος του ανηλίκου και του παιδιού σε όλες τις δραστηριότητες και φέτος έχουμε ένα εγχειρίδιο ε, για τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα, όχι μόνο για τα αεροδρόμια και τώρα το δοκιμάζουμε και στην επιχείρηση Θέμης. Ε, για το θέμα της διάστασης του φύλου και πώς ενσωματώνεται αυτό στις προσπάθειες. Ζητούμε ε, όλο και περισσότερο να έχουμε γυναίκες υπαλλήλου που να έχουν εκπαιδευτεί ειδικά σε αυτά τα θέματα φύλου που αφορά τη διακίνηση γυναικών, το τράφικινγκ και όχι μόνο. Αλλά είμαστε σε στενή συνεργασία με τον εκτελεστικό διευθυντή για να ενταχθεί και στο επιχειρησιακό σχέλος αυτή η πρόταση. Το Συμβουλευτικό Φόρουμ επίσης έχει πολύ μεγάλη δράση αναπτύξει το συγκεκριμένο τομέα. Είμαστε τώρα στο τελικό στάδιο για κατευθυντήριες γραμμές για τη δακτυλοσκόπηση. Έχουμε αρχίσει να συζητούμε με τους ε, υπαλλήλου σε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση ε, για το αν είναι κάποιος ανήλικος να χαρακτηρίζεται ανήλικος όταν υπάρχει ε, κάποια αμφισβήτηση. Ή στο θέμα ακόμα της δακτυλοσκόπησης έχουμε ζητήσει να είναι του ιδίου φύλου υπάλληλος γιατί υπάρχουν κάποιοι λαοί, κάποιες κουλτούρες που δεν, δεν σε αφήνουν καν να πιάσει το χέρι αν είναι από άλλο φύλο. Επίσης για τις μητέρες, τις Έχουμε για τις ε, αναγκαστικές επιστροφές ε, Έχουμε προχωρήσει επίσης από τις αρχές ε, της επιχείρησης και του νέου κανονισμού Έχουμε πάνω από 150 εκθέσεις και έχω και ήδη ε, προσωπική πείρα σχετικά με αυτά. Και έχουμε τρία βασικά συμπεράσματα. Σημαντικά θέματα ε, στις επιστροφές είναι τα ιατρικά. Ε, θέλουν οι ελεγκτές να έχουν να υπάρχει ένα υποχρεωτικό έγγραφο που να πιστοποιεί ότι για λόγους υγείας μπορεί να ταξιδέψει με πτήση ε, ε, ο ενδιαφερόμενος, γιατί μπορεί να υπάρχουν παθήσεις άγνωστες. Επίσης, η συνόδευτη ανήλικη είναι ειδικό κεφάλαιο για τη Frontex ε, στα πλαίσια της εγγύησης του, του, του συμφέροντος του ανηλίκου. Είναι πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο το θέμα αυτό. Και το τρίτο τώρα θέμα είναι η ειδική εστίαση στην επιχείρηση Focus, ε, και θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια θετικά η ταυτοποίηση και αναφορά ευάλωτων ομάδων συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν ειδικέ διαδικασίες στα hot για τους ανηλίκους, για τους αιτούντες άσυλο, για τα θύματα του τράφικινγκ. Όλα αυτά τα εξηγούμε στα σχέδια. τα ε, ανήλικα ε, παιδιά που είναι συνόδευτα και ε, κινδυνεύουν είναι μια ειδική κατηγορία και συμμετέχει και υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο στο ε, εγχειρίδιο. Και συμφωνώ με τον εκτελεστικό διευθυντή. Υποστήριξη ε, στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι βεβαίως επιχειρησιακός στόχος ε, των διαφόρων επιχειρήσεων του Frontex. Ακούσατε ήδη τις απόψεις του εκτελεστικού διευθυντή. έχουμε ενισχύσει ε, στην καταγραφή και στον έλεγχο ότι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στη δακτυλοσκόπηση επίσης. Επίσης χρειαζόμαστε μεσολαβητές, διερμηνείς κτλ. Αλλά η δακτυλοσκόπηση είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην αρχή πριν οποιαδήποτε άλλη. Και επίσης ε, δεν προβλέπεται παράδοση σε αρχές τρίτων χωρών, ούτε ε, αποβίβαση, ε, ούτε σύλληψη. Επίσης, επειδή υπάρχουν διάφορες ε, περιοχές αποβίβασης και διάφορα κέντρα καταγραφής ε, hot spot δεν είναι πάντα σαφές ε, σε ποια αρχή θα πρέπει να διαβιβάζεται η καταγγελία. Συνεργαζόμαστε πάντα με τις κατατόπους αστυνομικές αρχές που ασχολούνται με τα θέματα. Το τράφικινγκ διακίνηση ανθρώπων παραμένει αλλά δεν ανοιχνεύεται είναι σε πολύ διακριτικά επίπεδα. Χρειάζεται περισσότερη συνειδητοποίηση, περισσότερος ε, έλεγχος και κατάρτισης. Πάντως χρειάζεται στην πράξη μεγαλύτερη ενασχόληση με το θέμα. Άλλο πρόβλημα, η πρόκληση είναι οι αποβιβάσεις εκτός των hot spots, ε, των κέντρων καταγραφής και υποδοχής, που περισσότεροι αποβιβάσεις γίνονται εκτός των hot spot και χρειάζεται και, μέχρι και ιατρική ε, βοήθεια, παρακολούθηση, περίθαλψη. Όλα αυτά γίνονται με τρόπο λιγότερο διαθρωμένο από ό,τι στο hot spot. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν αποβιβάζονται, ε, οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν, δεν ενημερώνονται αρκετά για τις διαδικασίες ασύλου. Επίσης, στενή συνεργασία έχουμε επιδιώξει σε νέες δραστηριότητες προαναχωρησιακές παρατηρητές ε, αποστολές τρίτων χωρών ε, ταυτοποίηση, ταξιδιωτικά έγγραφα. Αυτό μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί η διεθνής προστασία. Παρακαλώ να συντομεύετε γιατί έχουμε ε, ε, καθυστερήσει. Και στους ασυνόδευτους ανηλίκους επιμένουμε πάρα πολύ υπάλληλοι να ε, ε, εκτιμούν ε, την ηλικία με τρόπο πάρα πολύ σοβαρό και όταν δεν είναι σαφής να προκρίνεται ότι είναι ανήλικος. Αυτά θα σταματήσω εδώ. Ναι, ναι, θα γίνουν και ερωτήσεις στη συνέχεια και στους δυο σας δεν έχουμε χρόνο, λέει ο πρόεδρος. Ωραία. Ξέρετε ότι στις 11 και 4 έχουμε ψηφοφορίες. Δύο-τρία λεπτά έκαστος, αν μπορείτε. Η κυρία Μετσόλα. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον κύριο Λεζένη που ήρθε για τις παρουσιάσεις. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω, έχει γίνει όμως πολλή συζήτηση σε σχέση με την επιχείρηση της Frontex και πόσο αποκλίνει από τις προηγούμενες επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων και την Triton. Θα ήθελα μια διευκρίνηση σχέση με τα όσα μας είπατε μέχρι τώρα. Πρώτα απ' όλα το την περιοχή που καλύπτει η επιχείρηση. Πόσο περισσότερο βορεία, του χώρου που κάλυπτε η Τράιτον έχει κινηθεί τώρα η Frontex και για ποιο λόγο. Θέλουμε πιο πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή φέρνει καλύτερα αποτελέσματα για τη διάσωση ζωών αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο κοντά στις ακτές της Λιβύης προκειμένου να σωθούν περισσότερες ζωές. Γιατί να πάει στα διεθνή ύδατα. Δεύτερον, ε, στις ε, αποβιβάσεις. Ε, αυτές γίνονται σε ασφαλείς λιμένες, εξασφαλίζονται συνθήκες ασφάλειας ή μπορεί αυτό να εξαρτηθεί από το ποιο συντονίζει τις επιχειρήσεις, πώς δηλαδή αξιολογούνται οι κανόνες αυτοί που εφαρμόζονται και επίσης σε σχέση με την αύξηση των αφήξεων από την Λιβύη υπάρχει κάποια ε, αναμένονται αυξήσεις αυτών των αφήξεων. Ο κύριος Διαστημέρα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Λεζερή και την κυρία Φερνάντες. Εγώ ήμουν ε, μάρτυρας της, ε, των εγγενείων, ε, της εξέλιξης, της πραγματικής μεταμόρφωσης του οργανισμού Frontex, ε, οργανισμού για την συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. Φυσικά έχουμε ε, πολλές διοικητικές δομές με τη Frontex, τη Eurojust, την Europol και ούτω καθεξής. Ποιος είναι ο ακριβής ρόλος ε, του οργανισμού Frontex στα κέντρα καταγραφής, γιατί ε, κανονικά ερευνά διασώζει, διανέμει, μεταφέρει. Έχουμε όμως σύντοση πολλών οργανισμών, πώς διαχωρίζονται τα διάφορα καθήκοντα και αρμοδιότητες. Επίσης, δεν έχουμε μόνο διάσωση ανθρώπινων ζώων, έρευνα, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και λαθροδιακή διακίνηση, εμπορία ανθρώπων, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, παράνομη ελεία, τρομοκρατία, λαθρεμπόριο όπλων. Οπότε έχουμε μία ζώνη που εμπίπτει στις μυστικές πληροφορίες, οι πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών για την εγκληματικότητα. Ε, οπότε μετά αυτά που μας είπατε φαίνεται να είναι απεριόριστη η αρμοδιότητά σας. Σε σχέση με την Ευρωπόλ ε, που έχει την ε, επιχείρηση Μάρε, η δική σας ε, υπηρεσία πώ οριοθετείτε Μιλάμε για το νομικό πλαίσιο. Ποια είναι η νομική, βάση πέραν του κανονισμού για να μπείτε στα χωράφια της, των μυστικών πληροφοριών για την εγκληματικότητα. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Φυσικά θαυμάζω το έργο σας, αλλά έχω εύλογες ε, αφιβολίες και ελπίζω να μου τις διασκεδάσετε. Η κυρία Κέγγε. Ναι, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και εγώ τους δύο μιλητές μας. Ξέρουμε ότι οι δραστηριότητες έρευνα και διάσωσης και από αυτό που βλέπουμε και στην ταινία έχει πολύ μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων της ε, επιχείρησης Θέμης. Ωστόσο, ε, δεν είναι δυνατόν, όσο εξαπλωμένε και είναι αυτές οι δραστηριότητε να καλύψουν ολόκληρο το χώρο της Μεσογείου. Άλλωστε αυτό μας το αποδεικνύουν και, οι, ε, και τα στοιχεία που μας δώσατε. 23% των διαδικασιών έρευνας και διάσωση καλύπτεται. Ε, τα υπόλοιπε λοιπόν επιχειρήσεις διάσωσης, έρευνας και διάσωση, τι αναλαμβάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει με μεγάλη αυτοθυσία. Και έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης από μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε ποιες περιπτώσεις δεν, υπογραμμίζω, δεν υπάγονται στην έννοια, δεν εμπίπτουν στην έννοια της ε, ε, διευκόλυνσης παράτυπης μετανάστευσης. Και κάτι ακόμη έχω συγκεκριμένη ερώτηση για τον κύριο Λετζερή. Υπάρχει περίπτωση κατά την οποία, από ό,τι λένε δικές μου πληροφορίες δηλαδή, έχουν οι λιβικές αρχές παρεμποδίσει έρευνα και διάσωση και διάσωση. Και αυτό το λέω γιατί και η, η οργάνωση Open Arms μας έχει δώσει τέτοια στοιχεία. Ε, επίσης, όταν γίνεται διάσωση στη θάλασσα από τις λιβικές αρχές, ε, οι πρόσφυγες αυτοί την χάνουν αξιοπρεπούς μεταχείρισης. Γιατί έχουμε πληροφορίες ότι τους επιστρέφουν στη Λιβύη και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Το δικαίωμα στην ε, υγειονομική περίθαλψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μπορούμε να μιλήσουμε για εθνοψυχιατρική, ε, για τις περιπτώσεις των ανθρώπων αυτών. Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως την χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε την περίπτωση μιας γυναίκας η οποία προσπαθούσε να περάσει τα σύνορα σε ε, φάση εγκυμοσύνης 7 μηνών ε, δεν μπόρεσε να περάσει και έχασε τη ζωή της τελικά. Υπάρχουν λοιπόν κάποια μέτρα για τα άτομα ε, τα οποία ε, είναι ανήλικοι μη συνοδευόμενοι. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για να πέσουν θύματα εμπορίου οργάνων και αυτό δεν το καταγράφουν οι επίσημες εκθέσεις. Ευχαριστώ κυρία Στέβενς. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα κι εγώ να, δώσω, να, να αντιδράσω στα σχόλια και τα αριθμητικά στοιχεία που μας προσέφερε η Frontex. Μας λέτε ότι είναι λιγότεροι αυτοί που, την, ε, που περνούν από τη Βόρεια Αφρική στην Ευρώπη. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όμως ακόμα, ο τύπος έγραφε ότι η European Stability Initiative, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Σταθεροποίηση, ένα ευρωπαϊκό η σταθερότητα, ένα ευρωπαϊκό think tank, θεωρεί πως ε, είναι αυξητικές οι τάξεις με 17.537 πέρυσι ετούνται στο άσυλο μόνο στο Βέλγιο και ότι δεν είναι καθόλου μειωτικές ε, ε, οι τάσει αυτές συμπεριλαμβανομένων και των νησιών τη Ελλάδος στο δεύτερο εξάμεινο του 2017 ήρθαν διπλάσιοι πρόσφυγες από ότι μέσα στο προηγούμενο 18 μήνο. Στη Γαλλία, στη Γερμανία επίσης έχουν αυξηθεί ε, τα αιτήματα οι αιτήσει ασύλου που κατατίθενται. Ερωτώ λοιπόν, διαπιστώνεται αυξητική τάση στους τελευταίους μήνες. Και αν ναι, τότε προφανώς έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αυτό το Think Tank μάλιστα ε, έλεγε ότι ένα από τα προβλήματα στην Ελλάδα και την Ιταλία ήταν ότι δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τις διαδικασίες για την ε, χορήγηση του ασύλου αυτά τα κράτη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι είναι ακόμα πάρα πολύ εκείνοι που περιμένουν στις χώρες ε, τη χορήγηση ασύλου. Γιατί αν συμβαίνει αυτό, κάποια στιγμή θα χάσουν την υπομονή τους. αφού ξέρουν ότι οι αρχές δεν θα διεκπαιρεώσουν αρκετά γρήγορα την αίτησή τους και θα προσπαθήσουν να φυγαδευτούν από τη χώρα για να πάνε αλλού. Ε, αυτό το αντιμετωπίζουν οι αρχές της Ελλάδας και της Ιταλίας. Έχει τελειώσει αυτό το πρόβλημα, είναι αποτελεσματικές διαδικασίες πλέον. Επίσης, πόροι και πιστώσεις. Θέλω να, να ξέρω τι έγινε, γιατί εδώ έχουμε πολλά προβλήματα σχέση με του ευρωπαϊκούς πόρους. Ευχαριστώ κυρία Σπινέλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον κύριο Λετζέρη και την κυρία Φερνάνδες ιδιαίτερος ε, για τη δουλειά τη. Την κυρία Φερνάνδες ιδιαίτερος λοιπόν θέλω να τη ρωτήσω αν ε, έχει την εντύπωση ότι αρκούν οι πόροι ανθρώπινοι και ηλικοί που έχει στη διάθεσή της για το τεράστιο αυτό έργο το οποίο έχει αναλάβει. Και έχω κάποια ερωτηματικά επί της ουσίας για την ε, Λιβύη και την επιχείρηση Θέμης. Τη ζώνη του Σαχέλ στην ε, Λιβύη. Από ό,τι βλέπω, συγγνώμη, ζώνη ΣΑΡ στη Λιβύη, δεν βλέπω να υπάρχει, από ό,τι μου επιβεβαιώνεται άλλωστε και ε, επισήμως αλλά και ατύπως, από τη Διεθνή Οργάνωση ε, Θαλασσών. Δεν υπάρχουν λοιπόν οι προϋποθέσεις για το Search and Rescue, SAR, και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ζώνη έρευνας και διάσωσης η Λιβύη. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί η ζώνη έρευνας και διάσωσης έχει θεσπιστεί έτσι ώστε να περιοριστεί και η δυνατότητα ανάληψης δράσης από τις μη ε, ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ένα δεύτερο. Και το έθεσε ήδη η συνάδελφος κυρία Μετσόλα. Έχει να κάνει με τους κανόνες για την αποβίβαση και αν αυτή η αποβίβαση γίνεται σε places of safety, δηλαδή σε ασφαλείς τόπους, όπως ορίζει η Σύμβαση ε, Έρευνας και Διάσωσης ή σε ε, σημείο που ίσως να είναι το εγκύτερο ε, από το σημείο διάσωσης, αλλά αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά για το αν θα είναι και ασφαλές σημείο. Επίσης, δραστηριότητες τρίτων και εφέμης. Είχαμε 35 μίλια ε, βεληνικές για την επιχείρηση τρίτων για ένα διάστημα το 2015 επεκτάθη. Τώρα έχουμε πάει στα 24 μίλια, θαλάσσια μίλια. Και ερωτώ με, το, με τη θέτη, όταν ένα φουσκωτό, γιατί για φουσκωτά μιλάμε, δεν μιλάμε για κανονικά σκάφη, φτάσει στα 24 μίλια, που είναι ο χώρος της ε, ευθύνης των Ιταλικών αρχών, Πότε θα φτάσει λοιπόν ένα τέτοιο ε, φουσκωτό στα 24 μίλια από τις Ιταλικές ακτές, αφού ξέρουμε ότι βυθίζονται πολύ πριν να φτάσουν στη ζώνη ευθύνης ε, του Ιταλικού κράτους. Κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε. Έχω μερικές ερωτήσεις προς εκπροσώπους ε, της Frontex. Μας είπατε κύριε Διευθυντά ότι πάνω από 6.000 ε, παράτυποι μετανάστες ε, πέρασαν χωρίς να εντοπιστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν έχει μειωθεί η τρομοκρατική απειλή σχέση με πριν από μία διετία. Σήμερα το πρωί φτάνοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είδα πάλι στρατιώτες ενόπλους περιπολίες και αυτό με τρομάζει πραγματικά. Είναι σαν να βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, όχι σαν να ζούμε σε ειρηνική εποχή. Οπότε εσείς, ε, αυτός ο ειδικευμένο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τι προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθεί ο κίνδυνος, να περιοριστεί η τρομοκρατική απειλή, γιατί μας λέτε ότι έχει μείνει αμύωτη σε σχέση με την προηγούμενη διετία. Και υπάρχει και το θέμα της δημόσιας συζήτηση για τη μετανάστευση. Αλλά το θέμα είναι πώς θα εξουδετερώσουμε αυτή την απειλή. Να ε, σκοτώσουμε στα σπάργανα αυτές τις αιτίες, να τις ε, εξαρθρώσουμε. Πώς θα τα καταφέρουμε. Μιλήσετε για νέους μηχανισμούς. Αλλά Έχω μια ερώτηση προς την κυρία Φερνάνδες. Μας είπατε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ανάλυσης των καταγγελιών και των ε, αιτιάσεων. Πραγματικά τα έχω χαμένα λίγο. Είπατε ότι για να κληθεί παραδεκτή μια ε, καταγγελία θα πρέπει να περάσει από μια περίπλοκη διαδικασία παρόλο που υπάρχει και η δυνατότητα ε, στο διαδίκτυο υποβολής καταγγελίας. Αλλά από πάνω από 90 καταγγελίες, ε, μόνο 5 έχουν κριθεί παραδεκτές. Πολύ μικρό ποσοστό. Επίσης, ίσως ειδικευμένος οργανισμός, που ε, αναγνωρίζουμε τη σημασία του, ε, τι κάνει για να εξασφαλίσει και την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα μειώσουμε τον κίνδυνο. Γιατί δεν διαπιστώσατε μείωση της τρομοκρατικής απειλής και της απειλής στην ασφάλεια. Ο κύριος Φουρτασούν, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λεζερή. Στα προγράμματα της Frontex ε, στην, ε, στη Μεσόγειο περιλαμβάνει και την ε, ε αποπομπή των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων και μάλιστα 11 μη ε, κυβερνητικές οργανώσεις έχουν εγκαταλείψει μόνο μία έχει σε 350.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μας λένε Financial Times και έχω μερικές ερωτήσεις. Ε, δεν θέλετε να επιστρέψετε, είπατε, ε, μετανάστες στην ε, Λιβύη. Ε, τι θα γίνει όμως, έχουμε ε, πληροφορίες ότι έχουν ε, μεταπιβεβαστεί σε λιβικό σκάφος ε, και θα επιστρέψουν στη Λιβύη. Επίσης μιλήσατε για την ζώνη ερεύνας και διάσωσης της Λιβύης. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απέρριψε το αίτημα τέτοια ζώνης για τη Λιβύη. Στις, στα 73 ναυτικά μίλια, τι, σε ποια ζώνη βρίσκεται ένα σκάφος πέραν της Λιβύης. Επίση, το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για την λαθροδιακίνηση προβλέπει θα πρέπει να μην τη χάνουν δίωξη ε, σκάφη που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης θα πρέπει για να κατηγορούνται να έχουν, να έχουν ε, κέρδη. Νομίζω ότι με βάση την ε, νοσιακή δημοθεσία, επαφείται στην απόλυτη διακριτική ευχήρια των κρατών μελών. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το θέμα, γιατί μερικές φορές και ανθρωπιστικά σκάφη κατηγορούνται για λαθροδιακίνηση. Επίσης, ε, τρίτη ερώτηση επαναλαμβάνω την ερώτηση μιας προλαλή σα. Έχετε, κυρία Φέραντε τα απαραίτητα μέσα για να ανταπεξέλθετε στο έργο σας, γιατί αυτή ήταν μια ερώτηση που αναφέρθηκε από το έργο του Frontex. Προκύπτει έλλειψη πόρων και μέσων για να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιούρεκ. Σας ευχαριστώ. Εμένα με ε, ενδιαφέρει μια ε, πληροφορία που για δεύτερη φορά την ακούμε στην Επιτροπή ότι το, η μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών είναι μετανάστες από την Ισία αυτή τη φορά. Η δεύτερη σε ε, σημασία εθνικότητα και ευχαριστώ για την ενημέρωση αλλά φαίνεται από τις πληροφορίες αυτές ότι δεν είναι μόνο ε, πολίτες που προέρχονται από την Ισία, αλλά και την Ίση πολίτες. Μέχρι στιγμής την Ισία μας φερόταν σχετικά σταθερή χώρα, που σχετικά ανώδυνα πέρασε την, ε, με την Αραβική Άνοιξη από την δικτατορία σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Οπότε έχω δύο ερωτήσεις. Ποια είναι τα αίτια αυτής της μετανάστευσης ε, από την, την Ισία. Εσείς ε, πού εντοπίζετε αυτά τα αίτια. Και δεύτερον, πρόκειται για άτομα που απλώς διέρχονται από την Τινησία ε, ή πρόκειται και για την ίσους πολίτες. Μήπως υπάρχουν και στην ε, Τινησία κάποια κυκλώματα λαθροδιακίνησης, όπως υπάρχουν αντίστοιχα κυκλώματα λαθροδιακίνησης στη Λιβύη, σε άλλες χώρες, μας τώρα έχουν αναπτυχθεί και στην Τινησία. Ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Λετζέρη και την κυρία Φερνάντες ε, για, τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπανε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια πτυχή, πέραν των όσων είπαν και οι συνάδελφοι. Όταν ήρθε το, η επιχείρηση Θέμης από την Ιταλία τουλάχιστον θεωρήθηκε ένα βήμα πρόοδου σε σχέση με την πρόοδο που, με τις υποχρέσεις που είχε μέχρι τότε αναλάβει η Ιταλία για την διάσωση, έρευνα και διάσωση στην ε, Μεσόγειο, αλλά και την υποχρέωση αποβίβασης μέχρι μεταφοράς και αποβίβασης στις Ιταλικές ακτές των διασωθέντων. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω μέσα σε αυτούς τους τελευταίους τρεις μήνες, δύο ουσιαστικά έτσι που έχετε ξεκινήσει, ε, ε πρόσφυγες έχουν υποδεχθεί χώρες άλλες πλην της Ιταλίας, γιατί ξέρουμε ότι έχουν μειωθεί οι αφήξει από τη Λιβύη, έχουν όμως αυξηθεί αφήξει από την Τινησία και άλλες χώρες και θα ήθελα να δω συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι η Ιταλία πάντα το, το, κράτο που, το κράτος που κατά κύριο λόγο υποδέχεται πρόσφυγες. Για την κυρία Στέβενες δηλαδή θα ήθελα να επισημάνω ότι 160.000 πρόσφυγες έχουν, μετανάστες έχουν φτάσει στην Ιταλία και είναι οι διαδικασίες της ε, καταχώρησης που έχουν επεκταθεί στο 100% για να καλύψουν το 100% των ε, ανθρώπων αυτών με, τις, ε, με την καταγραφή και δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ωστόσο το πρόβλημα πλέον είναι η υποδοχή και διαμονή των ανθρώπων αυτών και επιπλέον έχω να, σημειά να επισημάνω ότι έχουμε πλέον μετανάστες οι οποίοι φτάνουν από την ακτή του Ελεφανταστού, την Ερυθρέα και άλλες χώρες που δεν προβλέπεται ε, να μεταφερθούν σε άλλες χώρες. Θέλω λοιπόν να δω αν υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο υποδοχής και σχετική πρόβλεψη. Ένα άλλο ερώτημα, διότι και εγώ ανησυχώ ε, για το γεγονός ότι από το Δεκέμβριο οι αρχές της Λιβύης έχουν ε, λίγο πολύ παρετηθεί από την ε, υποβολή του αιτήματο ΣΑΡ ε, της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Θαλασσών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν υπάρχει έλεγχος αυτών των παράκτιων περιοχών, θαλασσιών περιοχών της Λιβύης και εάν αυτό σημαίνει ότι η αποβίβαση γίνεται όχι στην εγκύτερη τοποθεσία, αλλά στην ασφαλέστερη τοποθεσία, όπως ορίζει η σχετική σύμβαση, για τους μη συνοδευομένους ανελίκους. Εδώ και δύο χρόνια η Ιταλία έχει μια στοχευμένη προσέγγιση για την υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων οι οποίοι δεν ακολουθούν την πορεία και τους χώρους υποδοχής των υπόλοιπων ε, μεταναστών και προσφύγων αλλά έχουν ένα δικό τους δρομολόγιο στην υποδοχή των προσφύγων να ακολουθήσουν και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στις άλλες χώρες υποδοχής Μάλτα και Ελλάδα επί παραδείγματι ακολουθούν λοιπόν οι χώρες αυτές με τη δική σας υποστήριξη κανόνες ε, που έχουν να κάνουν πάνω απ' όλα με το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών όπως ορίζονται και στις Εθνικές συμβάσεις. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Έχουμε αρκετό χρόνο για τις απαντήσεις για αλλαγή. Να προσθέσω κι εγώ ή μάλλον να προτείνω να απαντήσετε πρώτα εσείς ε, κύριε Λεζερή και μετά κύριε Φερνάνδης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις για το που γίνονται οι αποβιβάσεις στα πλαίσια της επιχείρησης Θέμης. Ε, η επιχειρησιακή ε, ζώνη, επικράτεια της επιχείρησης Θέμης συμφωνήθηκε με τις Ιταλικές αρχές. Αυτό είναι ο κανόνας εκ του κανονισμού μας. Και κατόπιν ετήματος των Ιταλικών αρχών η επιχειρησιακή εμβέλεια ε, της επιχείρησης θέμης δεν επικαλύπτεται ε, με άλλες και, και περιορίζεται στην περιοχή έρευνας και διάσωσης που έχει ε, δηλώσει η Ιταλία. Οι κανόνες είναι σαφείς. Εφαρμόζουμε το Διεθνές Δίκαιο για την Έρευνα και τη Διάσωση και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι ο κανονισμός 65 του 2014 για τις επιχειρήσεις του Frontex που διέπει τις επιχειρήσεις εκεί και επίση υπάρχουν και διατάξεις από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θαλάσσης για τις αποβιβάσεις. Θα πρέπει και πάλι να επαναλάβουμε ότι δεν υπάρχει καμία αποβίβαση σε μη ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε στη Λιβύη, ούτε στην Τινησία, ούτε σε καμία άλλη χώρα της περιοχής που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί, συντονιστικοί μηχανισμοί για τα κέντρα ε, συντονισμού θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης. Και υπάρχουν και σύνδεσμοι ε, από τα γειτονικά κράτη-μέλη ε, στο, στη Ρώμη, στο ICC που είναι το κέντρο ελέγχου των επιχειρήσεων της επιχείρησης Θέμης. Έτσι ώστε τεχνικά να διευκολύνεται μια ομαλή ανταλλαγή υπηρεσιών και συνεννόηση όλων των ε, επιχειρήσεων και των δρόντων εκεί. περιμένουμε αύξηση ή μείωση των αφήξεων στη Λιβύη. Τι έχουμε διαπιστώσει από το θέρος του 2017. Υπήρξε μεγάλη μείωση των αφήξεων μεταναστών, 60% λιγότερες και από τις αρχές του έτους 70% λιγότερες αφήξεις από τη Λιβύη απευθεία. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις για το κέντρο καταγραφής hot spot ε, και κάποια νομικά ερωτήματα θέσατε για το Frontex και ε, τα διάφορα καθήκοντα που ε, εκτελούμε. Δεν έχει αλλάξει η έννοια του hot spot, του κέντρου καταγραφής και υποδοχής. Παραμένει έτσι όπως έχει σχεδιαστεί από το 2015 για την Ελλάδα και την Ιταλία. Δεν είναι διοικητική δομή, ε, ε, είναι μια επιχειρησιακή συνεργασία. Κάτι λέει ο κ. Διασδεμέρα εκτός μικροφώνου. Μα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς αυτό δήλωσε, ότι είναι διοικητική δομή. Εδώ, σε τούτη εδώ την Επιτροπή. Και βέβαια είναι διοικητική δομή. Εγώ είμαι πιο επιχειρησιακός. Εμείς δουλεύουμε εκεί επί τόπου και βλέπω ότι ο καθένας εργάζεται στα πλαίσια της εντολής του. Φυσικά υπάρχει ένας συντονισμός όμως των δραστηριοτήτων μας. Ο ρόλος του Frontex έχει ως εξή. Εμείς έχουμε δραστηριότητες φύλαξη των συνόρων, ε, ε, στα θαλάσσια σύνορα συχνά αυτό καταλήγει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σε τέτοια επιχείρηση ε, το πρόσταγμα έχουν οι αρμόδιες κρατικές αρχές. Μετατοπίζεται δηλαδή από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Μεταφορών ε, η ε, ευθύνη. Αυτή τη στιγμή αρχίζει μια επιχείρηση έρευνας και διάσωση, συντονίζεται από το Επιχειρησιακό Κέντρο στη Ρώμη και από το Ιταλικό Υπουργείο Μεταφορών πλέον και την Ιταλική Ακτοφυλακή. Τι σημαίνει αυτό. Ότι έχουμε υπαλλήλου του Frontex ε, ανεπτυγμένους που οφείλουν να, να ακολουθούν τους κανόνες και τις εντολές και τις οδηγίες που τους δίνει αυτό το Ιταλικό Κέντρο ε, Συντονισμού της Θαλάσσιας ε, Έρευνας και Διάσωσης. Οι διασωθέντες στη συνέχεια αποβιβάζονται. Αποβιβάζονται στα hot spots. Είναι γεγονός ότι καμιά φορά για λόγους χώρου αποβιβάζονται αλλού στην Ιταλία που δεν είναι επίσημα ε, κέντρα καταγραφής αλλά έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο η βοήθεια που παρέχουμε και η υποστήριξη ε, στις ταλικές αρχές. Ε, μπορούμε να βοηθήσουμε για την καταγραφή, για το screening, για την, ε, τις συνεντεύξεις με, με τους διασωθέντες, δακτυλοσκόπηση κτλ. Είναι υποστηρικτικό ο ρόλο μα προς τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και τι τοπικέ. Και το debriefing δηλαδή συζητούμε με τους ε, μετανάστες για να μάθουμε περισσότερα για την προέλευσή τους, την εθνικότητά τους, ε, τους λόγους που του οδήγησαν να ε, βρεθούν σε αυτό το σκάφο το οποίο διασώσαμε Και καμιά φορά έχουμε και κάποια προσωπικά δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κάποιες ε, έρευνες ε, ποινικές. Ε, εάν ο μετανάστης φαίνεται να έχει ανάγκη διεθνούς προστασίας, είναι ρόλος του υπαλλήλου Frontex να τους παραπέψει στις αρμόδιες αρχές για να κάνουν την αίτηση ασύλου. Αυτές οι αρχές μπορεί να είναι εθνικές ή και ε, συνάδελφοι του ΕΑΣΟ, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης Ασύλου. Εάν ανοιχνεύσουμε κάτι εμείς οι υπαλλήλοι μας που είναι ανισχυτικό ως προς την ασφάλεια, αν υπάρχει κάποια υποψία ότι ε, ο ενδιαφερόμενο μπορεί να εμπλέκεται σε αξιόπινες πράξεις διακίνηση και μεταναστών ή μπορεί να έχει ένα τρομοκρατικό υπόβαθρο ιστορικό, τότε αυτοί παραδίδονται σε για να γίνουν έλεγχοι δεύτερης γραμμή ε, ονομαζόμενοι από ε, την Ευρωπόλη ή τις Εθνικές Αστυνομίες. Νομική βάση γι' αυτό υπάρχει και είναι σαφή. Εμείς είμαστε οργανισμός αρμόδιος για τη φύλαξη των συνόρων και των ακτών για την καταπολέμηση ε, στα εξωτερικά σύνορα των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Έχουμε τέτοια εντολή και επίση έχουμε εντολή να συμβάλλουμε στην πρόληψη τη τρομοκρατίας πάντα σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά σύνορα. Δεν είμαστε υπηρεσία πληροφοριών ούτε αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ε, πάντα θα πρέπει να αναφέρουμε στην ε, Ευρωπόλ και στις εθνικές αστυνομίες και να παραπέμπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ε, τους ενδιαφερμένους. Τώρα, η εξεργασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων ε, επιτρέπεται, μας έχει δώσει την άδεια ο επόπτης προσωπικών δεδομένων. Το 2016 έγινε ένα πιλωτικό πρόγραμμα με την έγκριση του επόπτη για τα προσωπικά δεδομένα. Και όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα μας εντολή και συντονίσαμε το, η συνεργασία μας με τη Europol και τις Εθνικές Αστυνομικές Αρχές, ε, σημαίνει ότι κοινοποιούμε, εμείς δηλαδή, στον επόπτη προσωπικών δεδομένων, αντίστοιχο δικό μα αρμόδιο για τα προσωπικά δεδομένα και όλα αυτά με ε, άδεια του επόπτη Και λόγω της εντολής μας που τώρα ε, περισσότερο στρέφεται προς ε, δραστηριότητες επιβολής του νόμου και ε, τα προσωπικά δεδομένα, αποφάσισα να δημιουργήσω μία μονάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Έχω ένα μόνιμο υπάλληλο που ασχολείται με αυτά τα θέματα αποκλειστικά, γιατί όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα στον οργανισμό μας. Άλλες ερωτήσεις αφορούσαν την επιχείρηση Θέμης και το γεγονός ότι δεν καλύπτει όλη τη Μεσόγειο χωρικά. Η κατάσταση στη Λιβύη δεν είναι και πάρα πολύ ρόδινη, για να το πω έτσι. Στη Μεσόγειο τι έχουμε. Τρεις επιχειρήσεις ε, που έχει αναπτύξει ο Frontex. Η επιχείρηση Θέμης, που φιλοξενεί η Ιταλία, Έχουμε ακόμα το Ποσειδόν που φιλοξενείται στην Ελλάδα και την επιχείρηση Ίνταλο, μόνιμη επιχείρηση, την οποία φιλοξενεί η Ισπανία. Παλαιότερα αυτή ήταν εποχιακή, μόνο το καλοκαίρι. Αλλά ακριβώ λόγω των αριθμών και των στοιχείων και μετά για απαντώ και σε μια ερώτηση που έγινε για τις αφήξεις σε άλλα κράτη-μέλη. Προς το παρόν, η Ιταλία παραμένει το υπαριθμό ένα κράτος μέλος της αφήξης μεταναστών. Στη συνέχεια ακολουθεί, ακολουθούσε πέρσι η Ελλάδα ως δεύτερη και η Ισπανία ήταν στην τρίτη θέση. Οφείλω να πω ότι ε, αυξάνεται ε, κατά πολύ ε, ε, ο αριθμό των αφήξεων στην Ισπανία και μετά από συνεννόηση με τις Ισπανικές αρχές ε, αποφάσισα να είναι μόνιμη και η επιχείρηση Ίνταλο στην Ισπανία και όχι εποχιακή. Άρα συντονίζουμε τις δράσεις μας. Βέβαια με όλα τα μέλη υπάρχει και το Eurosur και όσο μπορούμε προσπαθούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, να μοιραζόμαστε πληροφορίες για επιχειρήσει έρευνα και διάσωση ή κατόπου που μπορεί να ενδιαφέρει τα κρατήρια. Ακόμα και είναι εκτό του δικού μα επιχειρησιακού χώρου. Η κατι αλλο που μπορει να ενδιαφερει τα κρατη μελη ακομα και ειναι εκτος του δικου μα επιχειρησιακου χωρου η κατασταση στη Λιβύη ε, τι να σας πω, εγώ μπορώ να σας πω ότι διαβάζω από τα δημόσια μέσα. Δεν έχουμε αναπτύξει εμεί επιχείρηση στη Λιβύη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεισφέρουμε στη δημιουργία ικανοτήτων στη Λιβύη και μέσα σε βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να είμαστε και μετριοπαθείς, γιατί είναι τεράστιο αυτό το εγχείρημα. Και όλοι ξέρουμε ότι οι συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στη Λιβύη δεν ανταποκρίνονται στις ανθρωπιστικές προδιαγραφές που θα περίμενε κανείς, που θα περιμέναμε εμείς από μια ευρωπαϊκή σκοπιά. Για τα στοιχεία τώρα των ετούντων άσυλου. Είναι αλήθεια ότι έχει αυξηθεί ο αριθμό αυτός. Για το ε, ε, παραμένει υψηλός ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου στα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι λίγο παράδοξο αυτό και το μελετούμε για να το κατανοήσουμε. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ο αριθμός των παράτυπων διαλέψεων σύνορων που ανοιχνεύονται στα εξωτερικά σύνορα μειώνεται. Σας είπα, ε, ε, πέρσι μειώθηκε κατά 60%. Παρ' όλα αυτά, ε, σε επίπεδο όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 60%. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη-μέλη δηλώνουν υψηλό αριθμό, αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων ασύλου. Αυτό εξηγείται με διάφορους τρόπους. Είτε ορισμένοι από εκείνους ήταν ήδη παρόντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ορισμένες αιτήσει από αυτές ε, οφείλονται σε δευτερογενείς μετακινήσεις από μία χώρα μέλος σε μία άλλη, Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και το γεγονός ότι περνούν απαρατήρητες κάποιες αφήξεις, γιατί είναι έτσι πιο αποσπασματικές, πιο κατακαιρματισμένες, είναι έσοδοι. Ε, ή μπορεί να είναι συνδυασμός όλων αυτών των αιτιών. Ε, ε, συνεργαζόμαστε με την ΕΣΟ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τα μελετήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Τέθηκε μία ερώτηση για το κατά πόσο και αφορά τον επιχειρησιακό μας χώρο, την επιχειρησιακή μας ζώνη. Ε, καταρχήν, ε, τα σκάφη που χρησιμοποιούν ε, οι μετανάστες και μερικές φορές είναι φουσκωτά και δεν φτάνουν στη διαδηλωμένη τελική ζώνη έρευνας και διάσωσης στην Ιταλική ΣΑΡ. Βέβαια, εμείς, σε ό,τι αφορά την έρευνα και διάσωση, η το δικό μας προσωπικό δεν επηρεάζεται από την επιχειρησιακή, δηλωμένη επιχειρησιακή ζώνη του Θέμης. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να παρέμβουμε σε περίπτωση λαθρεμπορίου ναρκωτικών εκτός ε, της δικής μας επιχειρησιακής ζώνης. Όταν όμως ε, μιλάμε για έρευνα και διάσωση, από τη στιγμή που υπάρχει ένα ε, κέντρο συντονισμού διάσωσης στη θάλασσα και που ενεργοποιεί το σύστημα και το δικό μας προσωπικό, μπορούμε καλύτερα να μεταβούμε στην περιοχή και να αναλάβουμε τα καθήκοντά μας, να διενεργήσουμε δηλαδή την έρευνα και διάσωση και μπορούμε να διασώσουμε τους μετανάστες και να τους φέρουμε σε ασφαλή λιμένα. Και με βάση τον κανονισμό 656 του 2014 ή με βάση το διεθνές δίκαιο αν ε, η επιχείρηση διάσωσης ε, δεν ε, εξασφαλίζεται ο συντονισμός της από το κράτος υποδοχής, από την Ιταλία για παράδειγμα, αλλά από άλλο κράτος μέλος, σε τέτοια περίπτωση θα υπακούσουμε στο συντονιστικό κέντρο και θα, μεταβούμε, θα κάνουμε την αποβίβαση εκεί που μας ε, υποδεικνύει το κέντρο συντονισμού να την πραγματοποιήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τρομοκρατικές απειλές, καταρχήν δεν είμαστε οργανισμός που ειδικεύεται σε θέματα τρομοκρατικών απειλών. Είμαστε οργανισμός συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Έχουμε ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων. Αλλά σε ό,τι αφορά τα αίτια της τρομοκρατίας, τι να σας πω. Σίγουρα είναι πολύ άριθμα αυτά τα αίτια. Και μερικά είναι άσχετα με τη διαχείριση των συνόρων. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των συνόρων πάντως, εμείς βάζουμε τα δυνατά μας για να συμβάλλουμε στην ασφάλεια και να μην περάσουν απαρατήρητες ε, κάποιες διελεύσεις των συνόρων. Κάνατε ερωτήσει για το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των κατευθυντηριών γραμμών που καλό θα ήταν να δίνονται στα κράτη-μέλη. Υπάρχει διδοντολογικός κώδικας, κώδικας συμπεριφοράς που εκπονήθηκε από την Ιταλική κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2017. Από ό,τι ξέρω, Πολλοί, πολλές ΜΚΟ δέχτηκαν να υπογράψουν αυτό το κώδικα συμπεριφοράς και να συνεργαστούν με τις Ιταλικές Αρχές και άλλους ε, εμπλεκόμενους παράγοντες όπως το Frontex. Πριν από δύο χρόνια είχαμε παράδειγμα τέτοιου κώδικα συμπεριφοράς στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές. Αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς ε, λειτουργεί ως κατευθυντήριες γραμμές ε, που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ και των δημοσίων αρχών επιβολής του νόμου. Πώς θα μπορούσατε να επιταχύνετε για να αφήσουμε λίγο χρόνο και στην κυρία Φερνάντε και ακολουθούν ψηφοφόρειες. Ναι, σε ό,τι αφορά την Τινησία, οι περισσότεροι μετανάστες από την Τινησία, τουλάχιστον η μισή από αυτούς, είναι οι υπήκοοι. Αλλά έχουμε και πολλούς από την Υποσαχάριο Αφρική, που χρησιμοποιούν την Τινησία για να περάσουν. Και είχαμε κάποιο προβληματισμό ως προς την ασφάλεια. Και μάλιστα μεγάλες κυκλοφορίες ε, βρετανικές εφημερίδες ε, πριν από λίγο καιρό είχαν αποκαλύψει κάποια σχετικά στοιχεία. Τώρα, τι γίνεται μετά την καταγραφή στα hot spots, στα κέντρα καταγραφής. Μετά την καταγραφή στα hot spots, οι μετανάστες που είναι επιλέξιμοι για διεθνή προστασία αναμένεται να περάσουν, να, να δρομολογηθούν προς τη διαδικασία ασύλου. Και όσοι δεν είναι επιλέξιμοι, οι οικονομικοί μετανάστες για παράδειγμα, που, για τους οποίους δεν υπάρχει άλλος ανθρωπιστικός λόγος ή οικογενειακός λόγους για να λάβουν την άδεια παραμονής θα επιστραφούν στη χώρα προέλευσης, εφόσον φυσικά πρόκειται για ασφαλή για αυτούς χώρα. Αυτά πάνω κάτω. Ε, να και από την Ίμακουλάδα Φερνάντες ε, την ευκαιρία να απαντήσει. Ναι, και νομίζω ότι ήταν καλό που μπορέσατε να απαντήσετε μέσα στον χρόνο Σα Ευχαριστώ και παρακαλώ την κυρία Φερνάντε να λάβει το λόγο. Θα είμαι και εγώ σύντομη πρόεδρο όσο μπορώ. Το δικαίωμα για φροντίδα μέρημνα, εκπαίδευση, παρουσία διακινητών, χώροι υποδοχής και δραστηριότητες μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε προσωπικό ιατρικό Μένα, αλλά δεν είμαστε αρμόδιοι για παροχή ατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι θέμα του κράτους υποδοχής Βεβαίω και μας απασχολεί το θέμα κάνουμε στο δυνατόν περισσότερο συντονισμό και παρακολουθούμε τα θέματα αυτά για την ε, εγκυμοσύνη και τις γυναίκες που αποθούνται. Είναι ενδιαφέρον θέμα διότι έχει εμφανιστεί αρκετές φορές και θα το συζητήσουμε σε μια προσεχή αναθεώρηση για τις κατευθυντήριες γραμμές, ιδιαίτερα για αυτές τις καταστάσεις. Γιατί δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη προδιαγραφή ως προς την απόθεση εγκύων γυναικών θα πρέπει να βρούμε μια κατευθυντήρια γραμμή αποδεκτή ώστε να μην είναι υποχρεωτική η απόθεση. Επίσης θέματα εκπαίδευσης. Εμείς δεν τα διαχειριζόμαστε. Είμαστε παρόντες κανονικά σε μέρη τα οποία, στα οποία μπορεί να υπάρχουν μάλλον δεν είμαστε παρόντες σε μέρη στα οποία κανονικά θα εμφανιστούν οι, ε, οι συνοδευόμενοι ανήλικοι. Είμαστε στη διαδικασία της καταχώρησης με την υποστήριξη που προσφέρουμε σε αρχές για την καταχώρηση και ταυτοποίηση. Και εκεί βεβαίως έχει σημασία να μπορούμε να ε, περνάμε τα στοιχεία των ε, ανηλίκων αυτών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, χωρίς προβλήματα. Επίσης θα πρέπει να πούμε, όπως σωστά επισημάνθηκε, ότι ε, δεν έχουν παρεμποδιστεί μέχρι τώρα οι λαθροδιακινητές και βέβαια και το πρόβλημα της, ε, του εμπορίου οργάνων είναι ορατό και πραγματικό. Ε, επίσης, στο προσωπικό και τη, γενικά την υποστήριξη που έχουμε. Δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα όσο σας θέλαμε για να αναπτύξουμε το δυναμικό μας. Ε, χρειάστηκε να προσλάβουμε έναν υπάλληλο ε, με καθυστερήσεις και με προβλήματα και νομίζω ότι θα πρέπει ε, να πούμε ότι πρώτα έπρεπε η δική μας ιστορική διαδικασία να ξεκινήσει να λειτουργεί, να είναι πλήρης και μετά να ανοίξουμε προς τα έξω. Έχω υλικό μαζί μου, θα σας το αφήσω για να το μελετήσετε αν θέλετε γιατί θέλαμε πάνω απ' όλα να ολοκληρωθεί η εσωτερική οργάνωση και μετά να γίνει η συζήτηση. Βέβαια τα παράπονα, οι διαδικασίες ε, παραπώνων και διαμαρτυριών δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Και ως προς την υποστήριξη στους πόρους σε οικονομικό επίπεδο, Έχουμε αυτή τη στιγμή έξι μέλη στην ομάδα, συμπεριλαμβανομένης και μου. Έχουμε την ε, γραμματεία του Συμβουλευτικού Φόρουμ, που ασχολείται μόνο με το Φόρουμ. Έχουμε βοηθό για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τη δική μου τη γραμματεία και γενικά τη γραμματιακή υποστήριξη. Είμαστε έξι λοιπόν μόνο. Και για να σε προλάβω Φαμπρίς θα πω ότι τρεις ακόμη ε, γραμματείς αναμένεται να ενταχθούν στην ομάδα εφέτος ακόμη. Άρα θα είμαστε συνολικά εννέα. Αλλά φυσικά αυτό δεν αρκεί για την κάλυψη των όλο και περισσότερων καθηκόντων της ε, ομάδας που στόχο έχει να διασφαλίσει την ε, τήρηση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Κυρία Σπινέλη, είχατε κάτι συμπληρωματικό, έχετε καλυφθεί. Όχι, όχι, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι και στα γαλλικά. Για τον κύριο Λετζέρι μια στομία ερώτηση. Ίσως να μην άκουσα καλά, να μην πρόσεξα καλά την απαντήση σας, αλλά μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε ότι η ζώνη έρευνα και διάσωσης της Λιβύας δεν υφίσταται, γιατί εσείς την παρουσιάσατε σαν δεδομένη στην προκατακτική σας, στην αρχική σας παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ναι, θα απαντήσω στα γαλλικά, μια και η ερώτηση ήταν και στα γαλλικά και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν θεωρώ δεδομένη την ζώνη έρευνας και διάσωσης της Λιβύης. Όχι. Υπήρξε μονομερής δήλωση το καλοκαίρι του 2017 η οποία γέννησε, προξένησε μια κατάσταση την οποία δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Στην ζώνη αυτή διαπιστώνουμε ότι κάποιες φορές η ακτοφυλακή της Λιβύης προβαίνει σε διάσωση στη θάλασσα. Επιχειρησιακά όμως η Frontex με την Λιβική Ακτοφυλακή δεν έχει ε, συνεργασία για τη διάσωση αυτή τη θάλασσα. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το δεδομένο ή το οριστικό αυτό, η ζώνη έρευνα και διάσωση. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, όπως ξέρουμε, για την κατασκευή ενός κέντρου συντονισμού τη θαλάσσια διάσωση στην Τρίπολη της Λιβύης που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ιταλία συμμετέχει και συνεργάζεται χάρη και σε ευρωπαϊκά κονδύλια και έχει ζητήσει η Ιταλία να συμμετάσχει και η Frontex να συνεργαστεί δηλαδή με την Ιταλία προσφέροντας την τεχνογνωσία της στις ακτοφυλακές. Επίσης η, η Cuba Libya, η ε, αποστολή πολιτικής προστασίας έχει συμμετοχή σε αυτό, κάλυπτεται επίση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεζερή, κυρία Φερνάντες, αγαπητοί συνάδελφοι για τις ερωτήσεις σας. 11 και 4 αρχίζουν οι ψηφοφορίες. Colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Καθίστε παρακαλώ. Όσοι ήθιστε ηλεκτρονικά. Για να μην χτυπήσετε, περιμένω να καθίσετε με ηρεμία. And we will begin. I know some people... Και ξεκινάμε γιατί ξέρω ότι έχετε και αεροπλάνα και τρένα να πάρετε. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα. Ξεκινούμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτη ψηφοφορία. Σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή των Μεταφορών. Σκρίπεκ διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών συστημάτων διοδίων, διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για την μη καταβολή οδικών τελών, αναδιατύπωση 24 Μαΐου στην ε, Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή. Κύριε Σκρίπεκ, θέλετε το λόγο όχι. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ, έχετε όλοι καθίσει, είστε έτοιμοι να ψηφίσετε. Ε, κουρασμένοι είμαστε όλοι, έρχεται και το Πάσχα. Α, σας αρέσει να είμαι λίγο πιο αυστηρός, έτσι. Λοιπόν, αρχίζουμε την ψηφοφορία. Πέρασε. Όχι, δεν ε, κλείσαμε την ψηφοφορία, την κρατάμε ανοιχτή ακόμη. Παρακαλώ, καθίστε όμως. Ψηφίσατε όλοι. Δεν έχετε ψηφίσει όλοι. Ψηφίσατε όλοι τώρα. Πέρας και εγκρίνεται 23. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται 24 αρχής ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 25 αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Η 28 αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 33 Πέρας. Εγκρίνεται 24. 34, 35 και 36 μαζί. αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται 37 αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 39 αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 40 άρχεται. Πέρας. απερίφθη 41 υπέρ. Πέρας. Εγκρίνεται 42, έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 43, υπέρ. Ε, άρχεται. Πέρας. Και απεριφθεί. Συμβαστική πρώτη υπέρ. Πέρας. Εγκρίνεται. 59 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 60 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 62 Πέρας. Εγκρίνεται. Τιολογικές αναφορές υπαριθμών 1, αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Απεριφθεί. Αιτιολογική σκέψη, τροπολογία 6, υπέρ. Πέρας. εγκρίνεται τροπολογία 7 αρχή η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 8 αρχή η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 9 άρχεται πέρας εγκρίνεται 10 άρχεται πέρας εγκρίνεται 11 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 12 άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται 14 άρχεται. Πέρασε. Απεριφθεί. 15 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται 16. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 18 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 2. Άρχεται η ψηφορία. Πέρασε. 20. Εγκρίθηκε προηγούμενα. 20. Πέρασε. Απεριφθεί. 21 η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 63 αρχίζει πέρας εγκρίνεται 64 η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται τελική ψηφοφορία και ονομαστικά παρακαλώ. Αρχίζει. Εγκρίνεται λοιπόν 54 ψήφισαν 48 υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές και συγχαρητήρια στον συντάκτη. So, Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία αγαπητοί συνάδελφοι. στην έκθεση Στίβενς για την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας. Πριν ε, την ψηφοφορία, η κυρία Στίβενς, η συγγήτρια, θα ήθελα μια σύντομη παρέμβαση να κάνει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε μια πρόσφατη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ σας παρουσίασα την κατάσταση των πραγμάτων Κάνατε κάποιες ερωτήσεις ε, για τη νομική διένεξη ε, Συμβουλίου και Επιτροπής και τι πιστεύω. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη διατύπωση του Συμβουλίου γιατί τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συντρέχουσα αρμοδιότητα για την ασφάλεια. Εγώ συγκέντρωσα τις διάφορες πολιτικές ομάδες και αποφασίσαμε από κοινού να προσθέσουμε κάποιες νομικές ε, συμβουλές και συστάσεις ε, στο ψήφισμά μας και ελπίζω όλες οι πολιτικές ομάδες να συμφωνούν και να είναι έτοιμες να ψηφίσουν τώρα αυτό το σημαντικό κείμενο. Καλώς, σας περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται 47 υπέρ 5 κατά, χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Συγγετρία. Περνάμε στην δεύτερη έκθεση Stevens που αφορά την πρόταση απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Ένωση του πρόσθετου πρωτοκόλου που συμπληρώνει τη Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την πρόληψη τη τρομοκρατία είναι συναφές με το προηγούμενο σημείο, το 13. Τη τροπολογία 1, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται 2, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται τροπολογία 3, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Τροπολογία 4. Η τρία εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με 49 ψήφου υπέρ, 5 κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια και πάλι κυρία Στίβεν. Περνάμε τώρα στην υπαγωγή νέων ψυχοδραστικών ουσιών και μέτρα ελέγχου. Στι 8 Φεβρουαρίου το Συμβούλιο ε, ζήτησε διαβούλευση για 7 ψυχοτρόπε ουσίε. Η αρμόδια συγκέντρια 26 Φεβρουαρίου υπέβαλε το σχέδιο έκθεση μετά τη νέα Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 14 Μαρτίου για νέε ψυχοτρόπε ουσίε. Τέσσερι καλύπτονται από τη Σύμβαση και περιλαμβάνονται αυτόματα στον ορισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για, τα, για τι ψυχοτρόπε ουσίε προκειμένου να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο ναρκωτικών δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε εκτελεστική απόφαση για αυτά τα νέε πέντε ψυχοτρόπες ουσίες και μάλιστα σας έχουμε μεταβάσει και τις επιστολές του Συμβουλίου. Όμως για τις δύο υπόλοιπε ε, ουσίες θα πρέπει να ψηφίσουμε. Δεν ξέρω αν η συγκήτρια θα ήθελε το λόγο πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες. Συγγνώμη που ήμουν τόσο γρήγορο και λίγο επιθετικό, αλλά ελπίζω να μην σα τρόμαξα. Αν θέλατε το λόγο να τον ζητούσατε. Μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Πολύ ωραία. Η κυρία Μάιτε Παγασαρντοντού Αρουής είναι η συγγετριά μας. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με 53 ψήφους υπέρ, μια κατά και χωρίς αποχές. Χαρητήρια, κυρία Ρουής. Περνάμε στη δεύτερη υπόθεση, το 16 της ημερήσης διάταξης, δεύτερη ψυχοτρόπος ουσία και πάλι ονομαστική κλίση, ψηφοφορία άρχεται. Τέλος. εγκρίνεται με 52 ψήφους υπέρ, μία κατά και χωρίς αποχές. Μπράβο και πάλι στην κυρία Ρουίθ. Περνάμε στο 22 τώρα σημείο, αγαπητοί συνάδελφοι, που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και του υποψηφίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Επιτροπή Επιλογή για το διορισμό του Γενικού Εισαγγελέα. Ο κανονισμό για την σύσταση του Γραφείου Ευρωπαίου Εισαγγελέα, όπω γνωρίζετε, θετήθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο και προκειμένου να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 2020, ήδη έχει ξεκινήσει η προεργασία. Σε ό,τι αφορά την επιλογή ε, και διορισμό του Ευρωπαίου Αρχή Εισαγγελέα και των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, άρθρο 14.3, ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή προβλέπει μια, μια επιτροπή επιλογής που θα είναι τετραμελή με πρώην μέλη από το, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, πρώην μέλη εθνικά της Eurojust, μέλη ανώτατων δικαστηρίων, ε, υψηλόβαθμού ε, εισαγγελείς και αναγνωρισμένους επιφανείς δικηγόρους. Ε, στις 5 Μαρτίου οι συντονιστές επιλήθηκαν και με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του σχετικού κανονισμού έχουμε δεχθεί από τις ομάδες τους εξή υποψηφίους. Θα τους διαβάσω με αλφαβητική σειρά. Κάντιτο Κόντε Πουμπίδο, Ρασίντα Ντατή, Εύα Ζολή, Αντώνιο Μούρα, και Μάριους Βορνησιάνου. Έχετε λάβει το κατάλογο των προτινομένων υποψηφίων και έχετε λάβει και τα βιογραφικά τους. Οπότε θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, με μυστική μάλιστα ηλεκτρονική ψηφοφορία και θα ψηφίσουμε διαδοχικά τους υποψηφίους, τον ένα μετά τον άλλο, με την αλφαβητική σειρά όπως τους διάβαζα και όλα. Οπότε θα ήθελα παρακαλώ σε κάθε ψηφοφορία ψηφίσετε μόνο υπέρ ενό υποψηφίου και για τους υπόλοιπους τέσσερις μπορείτε να ψηφίζεται κατά οι αποχές, οπότε θα ανάψει το γαλάζιο φως. Ψηφίζουμε για ένα μόνο υποψήφιο τη φορά. Για ένα μόνο υποψήφιο μπορείτε να ψηφίσετε και για τους υπόλοιπους αποχή. Για να ε, θα πρέπει να το κάνετε ενεργά. Δηλαδή είτε να ψηφίσετε όλου για του υπόλοιπου που κανονικά θα ήταν ισοδύναμη αποχή. Αλλά επειδή είμαστε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, να είναι ρητή η αποχή. Δηλαδή ενεργή αποχή, όχι να τεκμέρεται. όλου του υπόλοιπου. μπορούμε να ψηφίζουμε μόνο ένα. Έτοιμοι όλοι, θα ανάψει τον μπλε φως. Να τους ξαναδιαβάσω, τους υποψηφίους. Θα διαβάσω το όνομα και εσείς θα ψηφίσετε. Θα ψηφίσουμε, είπαμε με αλφαβητική σειρά. Πρώτος είναι ο κύριος Κάντιντο Κόντε Πουμπίντο. Άρχεται η ψηφοφορία για τον υποψήφιο Κάντιντο Κόντε Πουμπίντο. Ψηφίσατε. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεν χρειάζεται να διαβάσω το αποτέλεσμα. Περνάμε στη δεύτερη υποψήφια, την κυρία Ρασίδα Ντατή. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote closed. Τέλος ψηφοφορίας. τρίτη υποψήφια, η κυρία Εύα Ζολή. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος. Τέταρτος υποψήφιος, ο κύριος Αντώνιο Μούρα. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος. Και περνάμε στον πέμπτο υποψήφιο, τον κύριο Μάριους Φορνιτσιάνο. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. read them out now. So, so I'll announce the, yes. the one. So the elected person... Μάλιστα. Εκλέγεται η κυρία Ρασίτα Ντατή. So we have now, we go to the... Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγήτρια τη έκθεση είναι η κυρία Σπινέλη και δεν ξέρω αν θέλει η συγγήτρια το λόγο πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Όχι, προτιμώ να μην πω τίποτα. Ο κύριο Δία Δεμέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να δηλώσω την απόρριψή μου, απόρριψη για ένα υπενιγμό που γίνεται κατά της Ισπανίας της χώρας μου στην αιτιολογική έκθεση. Την απορρίπτω ε, γιατί ε, ε, και στερείται και υποβάθρου και είναι και άδικη και ανυπόστατη. Εντάξει, το σημειώσαμε. προχωρούμε στην ψηφοφορία. Συμβαστική 1 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 92, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 93, ψηφ... ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 96. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 101. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 102. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 103. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 104. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 105, άρχισε ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 106 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 2 άρχισε η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 110 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 111 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Η 112 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ανθρωπολογία 113. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 119, άρχιε ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4, άρχιε ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 124. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 125. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 132 τροπολογία, άρχιτε ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 133. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 134. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 135. 135 παρακαλώ ψηφίσουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 136 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 15 της Επιτροπής Πολιτισμού αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 138. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 139. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η Συμβαστική 6. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 147. αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 148. αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 149 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 7 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 152 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 8 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 9 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 168 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 169. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 16 της Επιτροπής Πολιτισμού αρχίζει ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 12 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 178 αρχίζει ψηφοφορία. Closed. Εγκρίνεται. 182 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 193 αρχίζει ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 13 αρχίζει ψηφοφορία. εγκρινεται Εγκρίνεται. Συμβαστική 13α αρχής ψηφοφορία. Συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, 13α, καλά το είπα. Αρχής ψηφοφορία. Το μηχάνημα αργεί σήμερα. Έλα. Το μηχάνημα αυτό. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Α. Μα αυτή ψηφίσαμε τώρα. Α. Η 197. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρασε. Rejected. 200. Απορρίπτεται. 200. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 201 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 203 η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 204 η ψηφοφορία. Πέρας. Δεν κρίνεται. Παράγραφος 17 της Επιτροπής Πολιτισμού αρχίζει η ψηφοφόρια. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 212 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 214 αρχής ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 215 αρχής ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 216 αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Rejected. Απορρίπτεται. 219. Αρχίζει η ψηφοφορία. 219. Πέρας. Εγκρινέται. 220. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 221, η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 222, η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 223, η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 224 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 226 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 227 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορές, η τροπολογία 1, αρχίζει ψηφοφορία. Trying to let nothing distract me. is closed. Πέρας, εγκρίνεται. Η τροπολογία 2, άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3, άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 και 7 ταυτίζονται αυτές. Ε, ψηφίζουμε και τις δύο τροπολογίες. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 11 αρχή ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 12 αρχή ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 13 Αρχίζει η ψηφοφορία. Rejected. Απερίφθη 14. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη 15 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 16. Πέρας. Απερίφθη 17. Άρχεται. Πέρασε. Απερίφθη 18. Πέρασε. Εγκρίνεται 19. Άρχεται. Πέρασε. Απερίφθη. 21. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 22. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις συμβαστική 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26, αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 27. Πέρας. Εγκρίνεται 28, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 16, αρχή του Πέρας. Και εγκρίνεται 34, αρχή του Πέρας. Απερίφθη 37. Πέρας. Εγκρίνεται 38, άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται 40, άρχεται. Πέρασε. Απεριφθεί 41, άρχεται. Πέρας Εγκρίνεται 42 αρκετά. Πέρας. Εγκρίνεται 43 αρχιτά Πέρας. Εγκρίνεται 44 και 70 είναι ταυτόσιμες. έρχεται η ψηφοφορία. πέρας. εγκρίνονται 45 αρχής ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 46 αρχής ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 47 αρχίζει πέρας Εγκρίνεται 48. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται 49. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται 17. Συμβαστική 17. Αρχιτεί ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 55 άρχεται πέρας εγκρίνεται 56 άρχεται πέρας εγκρίνεται 57 άρχεται η πέρας εγκρίνεται 58 Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 18 συμβαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 63. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται 19, συμβαστική 19, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 67 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 68 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 20 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 21 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται η 78 Πέρασε. Εγκρίνεται η 80 Πέρασε εγκρίνεται 82 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται για τις ε, παραγράφους της ε, Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων ψηφίζουμε την υπαριθμόν 8 άρχεται πέρας εγκρίνεται 9 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 15 της Τζούρι. Πέρας εγκρίνεται 23 άρχεται. Πέρας εγκρίνεται για την Επιτροπή Πολιτισμού. Παράγραφος 6 και τροπολογία. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται 18. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται 22. Άρχεται. Πέρας. Και εγκρίνεται 23 της Επιτροπής Πολιτισμού. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ονομαστικά. Αρχίζει. Πέρας. 44 υπέρ, 3 κατά, Τέσσερις αποχές και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Κύριε Γιούρεκ, έχετε διαδικαστικό. Ναι. Θα ήθελα απλώς να δηλώσω την ε, γνώμη μειοψηφίας, την άποψη της μειοψηφίας. Yes, that's still recorded. Thank you. Εντάξει, το σημειώνουμε. Ευχαριστώ. Έτσι τέλειωσαν οι ψηφοφορίε μα και η συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι. Αν δεν έχετε τίποτα στα διάφορα, 9 Απριλίου η προσοχή μα συνεδρίαση. Πέρα τη συνεδριάσεω, καλό Πάσχα. Καλέ διακοπέ του Πάσχα. Καλέ διακοπέ γενικώ. Well Διακοπές που τις ε, αξίζετε αν είστε κουρασμένοι όπως και εγώ. Σας εύχομαι πολύ καλές διακοπές.